Ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, αν ε, και δεν ε, είναι πολύ εξήμων εδώ, θα πρότεινα να ξεκινήσουμε. Υπάρχουν κάποια διαδικαστικά θέματα που πρέπει να δούμε και να αντιμετωπίσουμε. Το πρώτο ουσιαστικό θέμα έχει προβλεφθεί για τις 9 και 20 και είναι τα σημεία 6 και 7. Δεν είναι ακόμη εδώ οι συγητέ. Ίσως θα πρέπει λοιπόν να διακόψουμε για λίγα λεπτά τη συνεδρίαση, αλλά θα έλεγα να ξεκινήσουμε αντιμετωπίζοντα πρώτα τα διαδικαστικά θέματα. Καταρχήν θα έχουμε εκείνη παρουσίαση από την Κομισιόν για τα σημεία 6 και 7 και θα ξεκινήσουμε με το σημείο 7 και κατόπιν θα περάσουμε στο σημείο 6. Το σημείο 7 είναι ψυχοτροπέ ψυχοτροπές ουσίες. Ο κύριος Ποτασίεβιτ είναι ο συγητή και το 6 αφορά τη διακίνηση ναρκωτικών. κυρία Τερέσα Χιμένε Μπεσερίλη συγήτρια. Καλημέρα κυρία συγήτρια. Αν ε, δεν υπάρχουν αντιρρήσει, μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερησία διάταξη. Στη συνέχεια θα ήθελα να εγκρίνετε τι ακόλουθε ε, συν τάσει των συντονιστών έχουμε δύο διορισμούς εισηγητών. Καταρχήν ο κύριος Σεντοία Λαμπάρτ, ελπίζω να προφέρω σωστά το όνομά του, προέρχεται από το ΕΛΚ για τον Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση ΙΤΡΕ και στη συνέχεια πάλι από το ΕΛΚ, εξελβώς που θα είναι εισηγητής για την έγκριση τύπου ε, για τα οχήματα και την τροποποιητική οδηγία. Τη επιτροπή ΣΥΜΚΟ. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για αυτούς τους διορισμούς. Ωραία, σα ευχαριστώ. Κατόπιν. Μια άλλη ανακοίνωση σε ό,τι αφορά το γλωσσικό καθεστώς για σήμερα. Δυστυχώ δεν υπάρχει διερμηνία στα φιλανδικά, εστονικά, μαλτέζικα και κροτικά. Ζητώ συγγνώμη και ελπίζω να παραμείνει εξαίρεση. Είχαμε πρόβλημα την τελευταία φορά. Φτάνουμε στο σημείο 4 της ημερησίας διάταξης. Μία υιοθέτηση διευθετικού για την έκθεση Δίας Ντεμέρα. για την τροποποίηση του κανονισμού 539-2001 σε σχέση με το κατάλογο τρίτων χωρών, υπήκοοι των οποίων υπόκειται στην υποχρέωση θεώρηση για τη διάλυση των εξωτερικών συνόρων και υπήκοοι των οποίων απαλλάσσεται την υποχρέωση αυτή. Καθώ ο κ. Δίστα Μέρα πήγε στην Ολομέλεια πριν να λάβει χώρα η αναθεώρηση των ε, γλωσσομαθονομικών θα πρέπει να ξαναγίνει αυτή η εξέταση. Η συνήθι διαδικασία είναι ότι το αποτέλεσμα των γλωσσομαθονομικών παρουσιάζεται με τη μορφή ενό διορθωτικού. Και όπω έχουμε κάνει και στο παρελθόν, θα θεωρηθεί εγκεκριμένο το διορθωτικό αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει μέχρι το τέλο τη συνεδρίας σα Και βλέπω να βλέπω και καταφατικά ο εισηγητή. Μπορούμε να συμφωνήσουμε λοιπόν. Περνάμε στο σημείο 5 της ημερικής διάταξης παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιας πρότασης κατάργησης της απόφασης του Συμβουλίου 2007 κάθετος 124 που σχετίζεται με ένα ειδικό πρόγραμμα που θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους. Δεν λέμε εδώ ποιο είναι το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Στον ημερωτικό σημείο οι συντονιστές αποφάσισαν να ακολουθήσουν την απλουστευμένη διαδικασία βάσει του κανόνα 46 παράγραφος 1 και θα δώσω τώρα το λόγο στην Κομισιόν για να παρουσιάσει εν συντομία την πρόταση αυτή. Νομίζω ότι είναι η κυρία Σαββάρη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Σαβαρή, ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομο. Πρόκειται για ένα διαδικοστικό σημείο. Το πρόγραμμα αφορά την ε, πρόληψη ε, και τι συνέπειε της τρομοκρατίας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που διήρκεσε για το 2007-2013 και θα δικατασταθεί στο ταμείο, από το Ταμείο Εσωτερική Ασφάλειας μέσω της αστυνομία για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Γιατί αυτή η συγκεκριμένη διαδικασία γιατί συνήθως καταργούνται τα προηγούμενα ταμεία από τα προγράμματα που ακολουθούν για την περίοδο 2014-2020. Πρόκειται για μια διτή νομική βάση που υποστηρίζει το πρόγραμμα αυτό, σχετίζεται με τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και με τη συνθήκη Ευρατόμ. Για το λόγο αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία, να έχουμε ομοφωνήσει στο Συμβούλιο και διαβούλευση με το Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να καταργήσουμε αυτό το μέσο με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε. Πρόκειται λοιπόν για ένα διαδικαστικό σημείο, δεν θα μακρηγορήσω. Αυτή η κατάργηση φυσικά δεν πρόκειται να διακυβεύσει τη διαχείριση των ε, σχεδίων που τρέχουν αυτή τη στιγμή μέχρι να ολοκληρωθούν, χρηματοδοτούνται από το σημερινό πρόγραμμα, στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, ευχαριστώ να σας απαντήσω. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε. Θέλει κάποιο συνάδελφο το λόγο τότε θα παρουσιάσουμε μια πρόταση έγκρισης αυτής της πρότασης. Ευχαριστώ κύριε Σαβάρη. Περνάμε τώρα, τώρα στην κοινή συζήτηση για τα σημεία 7 και 6 με αυτή τη σειρά. Σημείο 7, νέες ψυχοτροπές ουσίες. Ε, ο κύριος Γιάτσεκ Προτασίεβιτς είναι εισηγητής από το ΕΛΚ και έχουμε και τι τη διατάξει σχετικά με τα στοιχεία τη αντικειμενική υπόσταση των εγκλημάτων και τι ποινέ που ισχύουν στον τομέα τη παράνομη διακίνηση ναρκωτικών όσον αφορά τον ορισμό ναρκωτικών. Η κυρία Χιμένη Μπεσερίλη είναι συγγήτρια για αυτό το σημείο και καθώς ε, έχουμε κερδίσει λίγο χρόνο, όχι πάρα πολύ βέβαια, Επομένω, αν δεν έχετε αντίρρηση θα έλεγα να προχωρήσουμε χωρί διακοπή. Καταρχήν θα έχουμε μια παρουσίαση της Κομισιόν, κατόπιν θα ακούσουμε και τους δύο εισηγητές και τους σκιώδεις εισηγητές και οποιοδήποτε άλλο μέλος που θα ήθελε το λόγο εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Λατεκνούτσε. Ε, thank uh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη, σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μας δίνεται να παρουσιάσουμε την πρότασή μας για τις ψυχοτρόπες ουσίες. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρόταση και για την Επίτροπο Ρέντινγκ και για την ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Τις οι διαπραγματεύσεις έχουν αρχίσει στο Συμβούλιο. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με όλους τους συναδέλφους και είναι πολύ θετικό το ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη ορίσει Αν υπομονούμε λοιπόν να συνεργαστούμε με τον κύριο Ποτασιέβιτς και τον κύριο Χιμένες Πισερέλη. διότι η συνεργασία αυτή θα είναι καλή για τη δημιουργία συνεργειών. Είναι ένα πακέτο λοιπόν για τις νέες ψυχοτρόπες ουσίες και έχει δύο πτυχές. Θέλουμε εμείς να καταστεί δυνατό να οριστούν ως ε, επιβλαβή σε ορισμένε ουσίε σε όλη την επικράτεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να προβλεφθούν ε, ποινικέ κυρώσει εξαιτία κινδύνων υγεία που αυτέ προκαλούν και να διασφαλίσουμε την ε, <clears throat> ελεύθερη κίνηση των ψυχοτρόπων ουσιών για νόμιμη χρήση. Όσον αφορά την ε, διάθεση και χρήση των ουσιών αυτών, ε, να πω ότι είναι ε, μια τάση που ίσως είναι από τις πιο επικίνδυνες τάσεις που παρατηρούνται στη σκηνή των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά οι ουσίες είναι διαθέσιμες εύκολα και έχουν παρόμοιες έχουν παρόμοιες ε, επιδράσεις όπως ε, η κάναβη ή το LSD. Από την άλλη όμως ε, δεν συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των ουσιών της σύμβασης του ΕΕ για τις ναρκωτικές ουσίες. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε προβλέψει να δημιουργηθούν περιορισμοί και να εισαχθούν περιορισμοί. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των νέων ψυχοτρόπων ουσιών που έχουν εντοπιστεί στην Ευρώπη έχει αυξηθεί με ταχύτατους ρυθμούς. Πάνω από 300 ε, ουσίε έχουν ε, εντοπιστεί από το 1997. Αλλά οι εθνικές ε, ειδοποίησει έχουν τριπλασιαστεί από το 2009 μέχρι το 2012 από 24 στι 73 κάθε χρόνο και 80% των ουσιών αυτών έχουν εντοπιστεί σε πάνω από ένα κράτος μέλος. Ήδη φέτος, δύο νέες ψυχοτρόπες ουσίες έχουν απαγορευτεί και η Ευρωπόλ και, η, ε, και ο Εθνικός Οργανισμός Ναρκωτικών Ουσιών συντάσσουν εκθέσεις για τέσσερις ακόμα ουσίες. Οι ενδείξει που έχουμε σε γενικέ γραμμέ είναι ότι η χρήση αυτών των ουσιών αυξάνεται και μια πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου δείχνει ξεκάθαρα ότι οι νέοι ανάμεσα στα 15 και 24 έτη έχουν χρησιμοποιήσει νόμιμες ε, ουσίες σε 5% από τις ουσίες αυτές. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς θα θέλουμε, θέλουμε να αναλάβουμε δράση για να προστατεύσουμε ιδιαίτερα τους νέους από τους κινδύνους των επιβλαβών ναρκωτικών ουσιών. Στην πρότασή μας απευθυνόμαστε μόνο ε, στις ουσίες αυτές όσον αφορά την απόσυρσή τους από την αγορά. Ουσίες οι οποίες ε, παρουσιάζουν κινδύνους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τα κράτη-μέλη προβλέπεται να αναλάβουν κατάλληλη δράση. Ε, προτείνουμε η ευρωπαϊκή δράση να είναι έξυπνη και να μην θέτει σε κίνδυνο την νόμιμη χρήση των χημικών ουσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην παρεμποδίσει την έρευνα την βιομηχανική και εμπορική χρήση των ουσιών αυτών. Οι οικονομικοί μας εφορείς χρειάζονται ασφάλεια δικαίου, διότι περίπου το 1 πέμπτο από τις ψυχοτρόπες αυτές ουσίες έχουν απόλυτα νόμιμη χρήση είτε για ε, κτηνιατρική, είτε στην ιατρική είτε στην βιομηχανία. Και αυτό πρέπει να συνεχιστεί φυσικά έτσι ώστε να ε, διασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία στην αγορά για νόμιμη χρήση των ουσιών αυτών. Ψήφισαμε λοιπόν αυτό το πακέτο για τις ε, ψυχοτρόπες ε, ουσίες και αυτό απαρτίζεται από δύο μέρη. Καταρχάς μια πρόταση κανονισμού που βασίζεται στο άρθρο 114 της συνθήκης για την εσωτερική αγορά και μια πρόταση οδηγίας η οποία βασίζεται στο άρθρο 83 ποινικού δικαίου το οποίο υπόκειται στην ε, υφιστάμενη απόφαση πλαίσιο. Τώρα, το πακέτο αυτό, όπως είπα, έχει δύο ε, προτάσεις, παρότι μιλάμε για έναν ενιαίο μηχανισμό. Ίσως ε, θυμάστε από πρόσφατες συζητήσεις πως βρισκόμαστε σε στάδιο τριμερούς διαλόγου. Υπάρχει ένας κανονισμός και οδηγία για την κατάχρηση της αγοράς. Η συνθήκη της Λισαβόνας δεν επιτρέπει το συνδυασμό νομική βάση που βασίζεται σε ποινικό δίκαιο με διατάξει από άλλα ε, κεφάλαια τη συνθήκη, όπω για παράδειγμα τη ε, εσωτερική αγορά. Το πακέτο λοιπόν αυτό στο σύνολό του θα αντικαταστήσει η φυστάμενη νομοθεσία. Θα γίνει τρόπον την άλλη λύση Γι' αυτό λοιπόν και ίσως αναγνωρίζετε ορισμένα στοιχεία που υπάρχουν στον κανονισμό. Κάποια πράγματα δεν έχουν αλλάξει δηλαδή. Παρότι λοιπόν η απόφαση, η παλιά απόφαση για τις ψυχοτρόπες ουσίες έχει λειτουργήσει ομαλά, υπάρχουν ορισμένα μειονεκτήματα. Καταρχάς η διαδικασία είναι αρκετά αργή, διότι υπάρχει ένα κενό τουλάχιστον 24 μηνών από την στιγμή που αρχίζει μια διαδικασία απαγόρευση σε μια ουσία μέχρι ότου τα κράτη-μέλη να ψηφίσουν τη σχετική νομοθεσία στο Συμβούλιο. Επίσης, το εφιστάμενο μέσο δεν ε, διαθέτει κάποιον ε, συγκεκριμένο μηχανισμό για να επιτρέψει προσωρινές ε, εξαιρέσεις σε περίπτωση άμεσου κινδύνου. Έπειτα, το δεύτερο μειονέκτημα είναι ότι ο παρόν μηχανισμός βασίζεται σε ποινικέ κυρώσεις ή δεν προβλέπει τίποτα απολύτως. Είναι άσπρο ή μαύρο δηλαδή και γι' αυτό το πεδίο δράσης μας είναι περιορισμένο και δεν ε, έχουν ληφθεί λοιπόν μέτρα σε πολλές περιπτώσεις ε, καθόλου διότι δεν είναι σαφές εάν ο κίνδυνος ε, μιας ουσίας είναι υπαρκτός ή τουλάχιστον αρκετά υψηλός έτσι ώστε να εισαχθούν ποινικές κυρώσεις. Ο εφιστάμενος μηχανισμός επίσης δεν λαμβάνει υπόψη τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Όσο υπάρχουν παρεκκλήσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη εξαιτία ε, των εθνικών τους δράσεων, τα διαφορές αυτές ε, ανακράτως ε, μέλος μπορούν να οδηγήσουν σε παρεμπόδιση της ενόμιμης χρήσης των ουσιών αυτών. Τώρα, εμείς τι κάνουμε με αυτό το πακέτο για να αντιμετωπίσουμε και να ξεπεράσουμε τα μειονεκτήματα αυτά. Καταρχά, ε, στην προσέγγιση μα έχουμε χρησιμοποιήσει μερικά στοιχεία. Μία βελτίωση είναι ότι έχει αυξηθεί η ε, ταχύτητα αντίδραση. Και αυτό κάνει τη διαφορά πραγματικά, ιδιαίτερα στην περίπτωση που χρειάζονται επίγοντα μέτρα. Ε, προβλέπουμε λοιπόν πολύ πιο γρήγορη δράση, έτσι ώστε ορισμένε ουσίες να αποσυρθούν από την αγορά, ενώ η διαδικασία λήψη αποφάση έχει απλοποιηθεί. Επίσης, ε, με αυτόν τον τρόπο από τους 24 μήνες το διάστημα αντίδρασης θα μειωθεί στους 10. Με έναν κανονισμό τα μέτρα θα είναι άμεσα εφαρμόσιμα έτσι, δηλαδή θα αποφύγουμε να πρέπει να λάβουμε ένα σύνολο αποφάσεων και θα μειώσουμε επίσης και την ε, υφιστάμενη περίοδο μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία που είναι 12 μήνες και θα φροντίσουμε ε, με την πρόταση αυτή να λαμβάνονται μέτρα πάρα πολύ γρήγορα όσον αφορά την διάθεση στην αγορά. Επίσης προβλέπεται μια, ε, ένας μηχανισμός άμεσης ανταπόκρισης για άμεσους κινδύνους προς τη δημόσια υγεία. Σύμφωνα λοιπόν με τον νέο κανονισμό θα εισαγάγουμε ε, προσωρινά μέτρα διάρκειας ενός χρόνου απαγόρευσης μιας ουσίας ε, από την αγορά. Και αυτό θα συμβεί ενώ διεξάγεται η εκτίμηση αντικτύπου. Αυτές οι ουσίες λοιπόν κατά τη διάρκεια ε, της ε, διεξαγωγής εκτίμησης αντικτύπου δεν θα διατίθεται στην αγορά έτσι ώστε να μπορούν να εισαχθούν έκτακτα μέτρα. Έπειτα το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με την αναλογικότητα. Εμείς εδώ εισαγάγουμε μια πολύ πιο ευέλικτη προσέγγιση με διαβαθμισμένο τρόπο. Υπάρχουν τρία επίπεδα κινδύνου, σε αντίθεση με τα δύο που έχουμε τώρα, δηλαδή είτε μη δράση είτε δράση με εφαρμογή ποινικού δικαίου. Έτσι λοιπόν τώρα σε μια τέτοια περίπτωση, ενώ πριν ή δεν υπήρχε δράση ή υπήρχε δράση, τώρα μπορούμε να έχουμε και μία ε, μέση λύση όταν υπάρχει ένας ε, μέσος κίνδυνος. Κυρία Κνούτσεν, λέει η Πρόεδρος, θα, μπορούσα, ήθελα να σας στήσω να ολοκληρώσετε. Το τρίτο λοιπόν στοιχείο είναι ότι προσπαθούμε να προστατεύσουμε την νόμιμη χρήση στην εσωτερική αγορά. Όπως σας είπα, 20% περίπου ε, των ουσιών αυτών είναι νόμιμες και χρησιμοποιούνται για ιατρικούς, ε, εμπορικούς και βιομηχανικούς ε, σκοπούς. Θέλουμε λοιπόν να διευκολύνουμε και να επιτρέψουμε την ελεύθερη διακίνηση και κυκλοφορία των ουσιών αυτών για νόμιμη χρήση. Η πρότασή μας λοιπόν θα οδηγήσει σε ένα αποτελεσματικό νομικό μέσο και να σας πω δύο λόγια για τη δομή, διότι είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζετε. Γιατί λοιπόν έχουμε δύο προτάσεις. Ο ε, κανονισμός είναι ο κρεγονίος λήθος και δημιουργεί τους αναγκαίους μηχανισμούς για εκτίμηση κινδύνου, για, ε, για υποβολή εκθέσεων και τον ορισμό των κριτηρίων για περιορισμού σε διάθεση στην αγορά. Και πιστεύω πως ε, η οδηγία επίσης ε, συμπληρώνει τον κανονισμό, διότι εισαγάγει ένα μια στοχευμένη τροποποίηση του εφισταμένου πλαισίου. Έχουμε διαλέξει αυτή την στοχευμένη τροποποίηση αντί μιας γενικότερη τροποποίησης, διότι υπάρχει η ανάγκη να αντιδράσουμε γρήγορα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν ε, διατάξεις ποινικού δικαίου για ορισμένες ουσίες οι οποίες απαιτούν ε, άμεση δράση, διότι είναι επιβλαβείς. Αυτά λοιπόν ε, σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει η πρότασή μας. Εν συντομία και πιστεύω πως χρειαζόμαστε κοινού κανόνες γιατί αυτοί θα οδηγήσουν σε μια αποτελεσματική πρόταση και αποτελεσματική εξίσου ανταπόκριση. Μέχρι τώρα έχουμε τη στήριξη αρκετών ευρωβουλευτών ε, και της Επιτροπής ε, αυτής και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την Επιτροπή και με την Προεδρία έτσι ώστε να δρομολογηθεί η πρόταση με όσο το δυνατόν ταχύτερο τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποιος εκ μέρους της Λιθουανικής Προεδρίας που θα ήθελε να προσθέσει κάτι. Ο κύριος Αμαρτίνκες, θα σας ζητούσα να είστε περιεκτικός. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρότασή της που έχει στόχο να ενισχύσει τον τρόπο αντίδρασής μας για την αντιμετώπιση των ουσιών για να λαμβάνουν τα σχετικά μέτρα και να μας δίνεται η ευκαιρία να αφαιρούμε από την αγορά τις επικίνδυνες ουσίες. Είναι μεγάλη σημασία των νομικών αυτών διατάξεων. Το Συμβούλιο έχει αρχίσει να τις επεξεργάζεται. Σήμερα μάλιστα συνεδριάζει η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου, στη διάρκεια της οποίας θα αναλυθεί κατάρθρο η πρόταση. Θα επιδιώξουμε να προωθήσουμε την πρόταση και θα συνεργαστούμε μαζί σας επικοδομητικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει η Σοφία Εντφέλτ. Εισηγητές, Προτασίεβιτς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ επίσης την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξαντλητική ανάπτυξη της οδηγίας και του κανονισμού. Ως εισηγητής σημειώνω ότι είμαι ανοιχτό σε κάθε είδους παρατήρηση δική σας και ενθαρρύνω τους πάντες και τις πάσες όχι μόνο και οδησηγητές να συνεργαστούν μαζί μου. Η έκθεση, το σχέδιο έκθεσης δηλαδή θα πρέπει να φτάσει στη μετάφραση στις 11.12. Θα συζητηθεί στις 9 πρώτου του 14 στην Επιτροπή μας και μέχρι τις 15 πρώτου θα πρέπει να μπορούμε να καταθέσουμε τις τροπολογίες. Επί της ουσίας, το πρόβλημα των ψυχοτρόπων ουσιών είναι πιο έντονο σε ορισμένες χώρες μέλη, όπου δεν αλλάζει η κατάσταση. Στην Πολωνία περάσαμε πραγματική κρίση αυτών των ουσιών το 2011. Σε ορισμένες χώρες μέλη ακόμα δεν είχαν σημειωθεί αρνητικές επιδράσεις των ουσιών αυτών. Σήμερα η κατάσταση ήδη έχει αλλάξει και άλλες χώρες επηρεάζονται σημαντικά από, την, αυτές. Πρόκειται για τομέα ο οποίος αναπτύσσεται ταχύτατα σε πολλές χώρες μέλη και βλέπουμε όλο και περισσότερους, ε, περισσότερα θύματα να καταλήγουν στα νοσοκομεία ή και στα νεκροταφεία. Το παρατηρητήριο τοξικομανίας λέει ότι μία μόνη ψυχοτρόπα ουσία έχει προκαλέσει 24 θανάτους έως τώρα. Αν εξετάσουμε το μηχανισμό που ισχύει σήμερα, της έγκυρης προειδοποίησης δηλαδή, απόφαση του 2007, σύμφωνα με τον μηχανισμό αυτό μόνο μία ψυχοτρόπος ουσία ανακοινώθηκε πέρσι, ενώ υπάρχουν 73 συνολικά. Και αυτό σημαίνει ότι το φαινόμενο εντείνεται. Να τονίσω ακόμη ότι οι αναλύσεις νέων ψυχοτρόπων ουσιών δείχνουν ότι πρόκειται για συνθετικές ουσίες, χημικά συντεθειμένες δηλαδή, τις οποίες ε, παράγουν ειδικευμένα εργαστήρια και είναι πολύ παρόμοια σύνθεσή τους με, τις ε, παράνομες, με τα παράνομα ναρκωτικά. Το επικίνδυνο είναι ότι οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν ποιες είναι οι δόσεις. Βεβαίως η παραγωγή των ουσιών αυτών δεν ανακοινώνουν και τις δόσεις, δεν περιλαμβάνουν και τις δόσεις μέσα ε, στα πακέτα. Γνωρίζουμε βεβαίως αρκετά καλά τα παράνομα ναρκωτικά σήμερα. Επομένως και οι καταναλωτές γνωρίζουν λίγο πολύ ποιοι είναι οι κίνδυνοι που απορρέουν από τη χρήση τους, ενώ για τις ψυχοτρόπες ουσίες δεν συμβαίνει αυτό. Άρα θεωρώ ότι είναι τελικά και πιο επικίνδυνες για την ουσία. Για να κατανοήσει κανείς καλύτερα το φαινόμενο, θα πρέπει να σημειώσει ότι σε αυτές τις ψυχοτρόπες ουσίες περιλαμβάνονται καμιά φορά μόλιβδος, ε, υδράργυρος, ε, χρώματα, δηλαδή ε, χρωστικές ουσίες και ούτω καθεξής. Φανταστείτε λοιπόν τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία τέτοιων ουσιών. Ουσίες οι οποίες πλήττουν περισσότερο τις νέες και τους νέους Ευρωπαίους. 5% σήμερα των νέων έχουν δοκιμάσει τουλάχιστον μια φορά τέτοιες, από αυτές τις νέες δηλαδή ψυχοτρόπες ουσίες. Υπάρχουν μάλιστα χώρες μέλη όπως τη Λιθουανία, την Πολωνία ή την Ιρλανδία πολύ υψηλότερα ποσοστά. Σε ό,τι αφορά τώρα την πρόταση κανονισμού, η Κομισιόν προτείνει την νομική βάση του άρθρου 114, δηλαδή την ενιαία αγορά. Από την άποψη των νομικών υπηρεσιών, κρίνεται ως ο καλύτερος συμβιβασμός για να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός. Αναμένω όμως από την Κομισιόν να αναπτύξει λίγο περισσότερο την νομική αυτή βάση. Νομίζω ότι ο κανονισμός αποτελεί καλή λύση διότι όχι μόνο μειώνει τις σχετικές προθεσμίες, αλλά δίνει και τη δυνατότητα απαγόρευση της κυκλοφορίας με άμεσο αποτέλεσμα κάποιων ψυχοτρόπων ουσιών. Άρα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια μας. Σήμερα χρειάζονται τουλάχιστον δύο χρόνια για να απαγορευτεί η κυκλοφορία μιας ουσίας. Μετά από την ε, θέση ισχύ των νέων κανόνων θα μπορέσει να περιοριστεί η προθεσμία αυτή στους 10 μήνες και σε ιδιαίτερα βαριές περιπτώσεις θα μπορεί να γίνεται άμεσα η απαγόρευση με διάρκεια ενός έτους. Πρέπει βέβαια να εξηγήσουμε ακόμη και το άρθρο 4 που έχει επιπτώσεις στην αρμοδιότητα των χωρών μελών. Μπορούν οι χώρες μέλη να απαγορεύσουν την ε, κυκλοφορία της ουσίας και τι συμβαίνει εάν μια χώρα μέλος θέλει να επιβάλλει αυστηρότερους κανόνες από αυτούς που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης με ικανοποιεί το άρθρο 14 που επιτρέπει ορισμένες χρήσεις για εμπορικούς σκοπούς, αλλά πρέπει εκεί να διευκρινιστούν ορισμένα ερωτήματα σε ό,τι αφορά τις πωλήσει μέσω διαδικτύου των ουσιών αυτών. Εν τέλει θέλω να πω ότι στην Πολωνία, την χώρα μου δηλαδή, το 2011 αρχίσαμε τον αγώνα κατά των ουσιών αυτών, αγώνας ο οποίος οδήγησε στην πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας των ουσιών αυτών. Πολύ σύντομα όμως διαπιστώσαμε ότι χάρη στην ενιαία αγορά δεν αρκούν οι εθνικές διατάξεις, εξαιτία δηλαδή της ενιαίας αγοράς. Και ιδιαίτερα για τις πιο βαριές ουσίες δεν πρέπει να επιτρέψουμε αυτές οι ουσίες να μπορούν να πολλούνται σε όμορες χώρες εφόσον απαγορεύονται σε μία χώρα ή να αγοράζονται μέσω του διαδικτύου. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι και νέες ψυχοτρόπες ουσίες, οι νέες ψυχοτρόπες ουσίες έχουν χαμηλό κόστος παραγωγής. Μάλιστα, διάβασα και ένα άρθρο για το οργανωμένο έγκλημα. Μάλλον είναι ένα, με είναι ένα είδος που ενδιαφέρει ιδιαίτερα το οργανωμένο έγκλημα για τους λόγους αυτούς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Έχουμε κάποιο ε, χρόνο, διότι είχαμε προβλέψει μέχρι τις 10 την συζήτηση του θέματος αυτού. Απλώς παρακαλώ όλες και όλους να δείξετε κάποια αυτοσυγκράτηση και να είσαστε σύντομοι, γιατί αλλιώς θα ξεπεράσουμε τον χρόνο ήδη από την πρώτη συζήτηση. Γι' αυτό και σας παρακαλώ να είστε συντομότεροι. Χιμένες. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομη, γιατί πιστεύω ότι και η Κομισιόν αλλά και ο εισηγητής του κανονισμού ανέφεραν πολλά από τα στοιχεία, επομένως δεν θα επαναληφθώ εγώ εδώ. Και επίσης ε, σίγουρα θα ξανασυζητήσουμε το θέμα αυτό γιατί σήμερα απλώς έχουμε την παρουσίαση εδώ. Ευχαριστώ την Κομισιόν που μας παρουσιάζει την απόφαση τροποποίησης για την απόφαση πλαίσιο του 2004 σε σχέση με τη θέση ψηλέξεων διδάξεων σχετικά με τα στοιχεία αντικειμενική υποστέση των εγκλημάτων και τι ποινέ που ισχύουν για τη διακίνηση των ναρκωτικών. Επίση, οι νέε ψυχοτρόπε ουσίε έχουν εισαχθεί στην αγορά σε πολλά κράτη-μέλη και αυτά τα νέα ναρκωτικά είναι μεταξύ τη νομιμότητα και τη παρανομία και ζημιώνουν την υγεία των ατόμων και ιδίω των νέων. Επίσης, αυτές σχολούνται πολλές εγκληματικές οργανώσεις που θέλουν να παράξουν και να κυκλοφορήσουν αυτές τις ουσίες, σαν να ήταν νόμιμες ψυχοτρόπες ουσίες. Πρέπει λοιπόν να επικαιροποιήσουμε την νομοθεσία μας. Το πρόβλημα αυτό είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και πρέπει να καταπολεμηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο από ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. Μόνα του. τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν. επομένω είναι σκόπιμο αυτό το πακέτο που μα παρουσίασε η Κομισιόν ω εισηγήτρια αυτή της πρόταση. Ε, θα βελτιώσω στο μέτρο του δυνατού αυτό το κείμενο μαζί με του Σκιώδη, το Συμβούλιο, την Κομισιόν ε, και θα συνεργαστώ και με τον εισηγητή περί του κανονισμού. Και καθώς κάνουμε τώρα τα πρώτα βήματα για την ανάπτυξη αυτής της έκθεσης, θα ήθελα να θέσω δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις στην Κομισιόν. Στο αιτιολογικό, στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης αυτής, η Κομισιόν αναφέρεται στον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει αυτή η έκθεση στα θεμελιώδη δικαιώματα. Μπορείτε να μας πείτε σε τι ακριβώς αναφέρεστε, σε ποιον αντίκτυπο και δεύτερο, ποιο είναι το αποτέλεσμα της οδηγίας 2004 στην παράνομη τα πολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και πώς μπορούμε να τη βελτιώσουμε εδώ από το Κοινοβούλιο, γιατί βάσει όσων άκουσα, ε, στη συνεδρίαση που κάναμε για τις συνέπειες αυτών των ναρκωτικών, ποια είναι αυτά τα ναρκωτικά, να τα διαχωρίσουμε τα νόμιμα από τα παράνομα ναρκωτικά. Μπορώ να σας πω ότι δεν κατάλαβα πάρα πολύ καλά τι ακριβώς γίνεται με τη διακίνηση των ουσιών αυτών και ε, πώς μπορεί να επηρεάσει η συνεργασία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Σας ευχαριστώ. Θα ανοίξω το λόγο για τη συζήτηση. Έχω άτομα που έχουν ζητήσει το λόγο, ένα σκιώδη και δύο συναδέλφους, τέσσερις. Τώρα, άλλος κανείς. Κύρκοφ, Τριανταφυλλίδης, Ματιέ, και Ρεμπρόντς. Άλλος κανείς. Μάλιστα, κλείνω τον κατάλογο. Και θα σας ζητήσω να περιοριστείτε στα δύο λεπτά, Κύριο Σκέρκοφ. Ναι, μιλώ σκιώδης. Ήθελα να ξεκαθαρίσω, Πρόεδρε, ότι εδώ συμμερίζομαι τις ανησυχίες όλων για τα θέματα αυτά. Έχουμε χάσει πάρα πολλούς νέους στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της κατανάλωσης αυτών των ουσιών, ψυχοτρόπων ουσιών και πρόδρομων ουσιών. Νομίζω ότι είναι τραγική κατάσταση για την Ευρώπη. Εγώ συμμερίζομαι τις ανησυχίες της Κομισιόν για τον κίνδυνο ε, στην υγεία των Ευρωπαίων πολιτών και υποστηρίζουμε τις προσπάθειες του Διευθυντής Europol ε, να βελτιώσει τη χρήση της βάσης δεδομένου της Europol για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Είδαμε και την αξιολόγηση Κομισιόν ότι πρόταση κανονισμού και για οδηγία που να θέτει ελάχιστες διατάξεις για τα στοιχεία αντικειμενικής υπόστασης ε, των ε, εγκλημάτων και τις ποινέ. Εμείς θεωρούμε ότι εδώ θα πρέπει να αφαιθεί ε, στην αρμοδιότητα των κρατών μελών το θέμα των ποινών. Βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι σε καλύτερη θέση να περιορίσει τη διαθεσιμότητα αυτών των ουσιών στην ενιαία αγορά γιατί τα κράτη-μέλη δεν μπορούν ε, να αντιμετωπίσουν όπως πρέπει την κυκλοφορία αυτών των ουσιών. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Η διάδοση των νέων ψυχοτρόπων ουσιών επηρεάζεται από πάρα πολλού παράγοντε. Ε, έχουμε διεθνεί και εθνικέ και τοπικέ δυνάμει. Όλα αυτά εκδηλώνονται πολύ διαφορετικά στα διάφορα κράτη-μέλη και ο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία είναι διαφορετικό ακριβώς ανάλογα με την τοποθεσία. Έχουμε διαφορετικά συστήματα για να αντιμετωπίσουμε τα ναρκωτικά γενικά. Και εδώ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ευέλικτοι. Έτσι λοιπόν, αν και υπάρχει προσθέμενη αξία από την ευρωπαϊκή δράση, κυρίως ό,τι αφορά στην ανταλλαγή πληροφοριών και στην παροχή ανάλυσης από τη Europol και από άλλους, εγώ συμφωνώ, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι εδώ δεν θα χάσουμε τη δυνατότητα λήψη πρωτοβουλίας, ε, γιατί ε, ουσιαστικά το να αντλήσουμε πληροφορίες και πόρους και να κάνουμε μια προσπάθεια εκπαιδευτική είναι ο κύριος τρόπος για να σταματήσουμε ε, την, ε, το να πάνε αυτές οι ουσίες ε, στα λάθος χέρια. Κύριος Τρινταφυλλίδης. Πολύ σύντομα, κυρία Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν και τους συζητητές για το έργο τους. Φυσικά θα το εξετάσουμε πάρα πολύ προσεκτικά όλα αυτά. Εγώ θέλω να πω ότι η δική μας ομάδα είναι κάπως ε, σκεπτική στην υιοθέτηση των κανονισμών, αλλά σε ό,τι αφορά ε, το αντικείμενο θα διατυπώσουμε τη θέση μας βάσει όσων ακούσαμε σίγουρα σήμερα και θα συνεργαστούμε πολύ στενά με τους εισηγητές τις επόμενες συνεδριάσεις. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ήσασταν πάρα πολύ συνοπτικός. Η κυρία Ματιέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την πρότασή της γιατί είναι πραγματικά ανησυχητική η πραγματικότητα. Οι νέες ψυχοτρόπες ε, ουσίες ε, αυξάνονται, κάθε εβδομάδα κοινοποιείται κάθε Κάθε εβδομάδα κοινοποιείται μία νέα ουσία. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος επί των πωλήσεων, ούτε πληροφορούνται οι καταναλωτές. Και οι νέοι είναι οι κύριοι καταναλωτές και διατρέχουν πολύ μεγάλους κινδύνους. Το 5% των νέων στην Ευρώπη έχουν ήδη καταναλώσει αυτές τις ουσίες μία φορά στη ζωή τους. Ε, αυτές ε, οι ουσίες μπορεί να παρουσιάζονται με έναν τρόπο που να μην θεωρούνται θεωρούνται επικίνδυνες, όμως τελικά επιφέρουν πολύ μεγάλο κίνδυνο για την υγεία, πολύ μεγαλύτερο ίσως και από τα παραδοσιακά νοκορτικά. Πρόκειται για μια γκρίζα ζώνη και δεν ξέρουμε ακόμη τα αποτελέσματα των ουσιών αυτών και πόσο εθιστικές είναι. Θα πρέπει λοιπόν ε, να απαντήσουμε ώστε να τον καλύτερα στα προβλήματα της εξάρτησης και της τοξικομανίας. Θα πρέπει να γίνει μια ανάλυση κινδύνου και να εναρμονίσουμε τις απαιτήσει μας για τις παράνομε ουσίες. Και όπως είπαν πολλοί συνάδελφοι, το εμπόριό συνεχίζει να ε, τροφοδοτείται οι εγκληματικέ οργανώσεις ε, και φυσικά δεν υπάρχει οπαρκής έλεγχος και γι' αυτό είμαστε πολύ θετικοί απέναντι στην πρόταση της Κομισιόν και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να την υφετήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ κύριος Μπρόνς, τελευταίος ομιλητής. είπε εκπρόσωπος της Κομισιόν ότι ήθελε να αποτρέψει την παράνομη χρήση αλλά όχι την νόμιμη χρήση. Η νόμιμη χρήση θα μπορούσε να αφορά δύο κατηγορίες, την ιατρική χρήση ή μια βιομηχανική χρήση όμως δεν μας εξήγησε ίσως γιατί δεν είχε αρκετό χρόνο για το πώς θα γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα αν μιλάμε για κάτι που έχει μια νόμιμη ιατρική χρήση, τι θα συμβεί, θα χορηγείται μόνο από γιατρούς, θα γράφεται ως συνταγή ή θα αγοράζεται μόνο παρουσία των φαρμακοποιών και φυσικά έχουν διαφορετικές αρμοδιότητες οι φαρμακοποιοί ανάλογα με τη χώρα. Νομίζω ότι είπε εκπρόσωπος της Κομισιόν ότι θα συνοδευτεί ο κανονισμό και από οδηγία. Αυτέ οι λεπτομέρειε λοιπόν θα περιλαμβάνονται στην οδηγία και θα αφήνουν τα κράτη-μέλη ελεύθερα να αποφασίσουν για την επίτευξη του στόχου. Και φυσικά ένα συναφή μεγαλύτερο κινδύνο που μπορεί να καλύπτεται και από το επόμενο σημείο στην ημερησία διάταξη δεν είναι μόνο των αυτεντικών ουσιών ε, όπου έχουμε κατάχρηση και παράνομη χρήση, αλλά ίσω να έχουμε μία παρασκευή των ουσιών με ένα λανθασμένο τρόπο μπορεί να είναι ακόμη πιο επιζήμιες. Σας ευχαριστώ. Είχαμε δύο ερωτήσεις από την κυρία Χιμένες. Στέθηκαν στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Κυρία Κρούτσεν, μπορείτε να απαντήσετε. Ε, thank you. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ όλους τους ομιλητές για τη στήριξή τους και τα πολύ χρήσιμα σχόλιά τους. Ε, σημείωσα αρκετές ερωτήσεις. Μία από αυτές ε, αφορούσε τη νομική βάση της εσωτερικής αγοράς. Και πράγματι, αυτό είναι η καλύτερη και σωστότερη λύση, όπω είπε και ο εισηγητή, διότι αυτό που προσπαθούμε εμεί είναι να απαγορεύσουμε τι ε, βλαβερέ ουσίε από την αγορά, ενώ ταυτόχρονα να διευκολύνουμε την ελεύθερη κίνηση των ουσιών που έχουν νόμιμη χρήση. Η νομική βάση στην ε, ενιαία αγορά μα επιτρέπει να προστατεύουμε του καταναλωτέ και την υγεία του. Έχουμε λοιπόν ε, αυτόν τον διπλό στόχο και πιστεύω πως αυτή είναι κατάλληλη νομική βάση για αυτό. Τώρα, Όσον αφορά το διαδίκτυο, αν θυμάμαι καλά υπήρχε μια ερώτηση για το διαδίκτυο. Δεν αναφέρεται ε, σαφώς το διαδίκτυο στην πρόταση, αλλά να σας πω ότι καλύπτεται, διότι όλες, όλες οι δύο δι, ε, θα συμπεριληφθούν. Δεν υπάρχει λοιπόν ανάγκη για συγκεκριμένη αναφορά του διαδικτύου. Φυσικά και το έχουμε λάβει υπόψη αυτό. Τώρα, όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, καμία ερώτηση του κυρίου Χιμένες. Κυρίες. Η οδηγία αναφέρει στο επεξηγηματικό σημείωμα ότι ενδεχομένως υπάρχει μια έμεση, υπάρχουν έμεσες επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα, στο ποινικό δίκαιο δηλαδή τροποποιώντας το πλαίσιο. Αλλά στην ουσία δεν είναι τίποτα περισσότερο από αυτό που έχουμε ήδη τώρα. Δεν υπάρχει επέκταση ε, του ποινικού δικαίου δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σε σχέση με την νομοθεσία που έχουμε ήδη για τις ψυχοτρόπες ουσίες και φυσικά πρέπει να σημειώσουμε ότι οι κυρώσεις του ποινικού δικαίου δεν θα επεκτείνονται στους χρήστες. Δεν υπάρχει λοιπόν ε, άμεσο αντίκτυπος στους χρήστε. Οι ποινικέ κυρώσεις αφορούν τους προμηθευτέ, είτε ε, αυτέ ε, βρίσκονται στο εθνικό δίκαιο, είτε αφορούν συγκεκριμένους ε, μεμονωμένους χρήστες. Τώρα, αναφερθήκατε στο οργανωμένο έγκλημα. Πιστεύω πως ε, το κύριο σημείο είναι ότι ναι, η Ευρωπόλ ασχολείται από την αρχή με τη διαδικασία αυτή, είναι αναμειγμένη από την αρχή ε, στη διαδικασία, γίνονται ειδοποιήσεις, η Ευρωπόλ συνεργάζεται με, το, με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ναρκωτικών Ουσιών συνεργάζεται επίση με τα κράτη-μέλη. Υπάρχει μια ειδική επιστημονική επιτροπή όπου συγκεντρώνονται όλε οι πληροφορίε για το οργανωμένο έγκλημα, πληροφορίε και από την Ευρωπόλ και ε, συγκεκριμένα επιστημονικά στοιχεία. Πιστεύω λοιπόν ότι η Ευρωπόλη μπορεί να συμπεριλάβει τι πληροφορίε αυτέ στη στρατηγική τη για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Τώρα, όσον αφορά τι ε, δυνατότητε ε, δράση από τα κράτη-μέλη, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δράση θα λαμβάνεται μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μόνο για τις ουσίες οι οποίες έχουν ε, κινδύνους για όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επίσης σημαντικό να υπάρχει μια εκτίμηση κινδύνου για τον συνολικό αντίκτυπο μιας ουσίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει. Τώρα, αυτέ οι 300 ειδοποιήσει που έχουμε μέχρι τώρα, να σα πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει προ το παρόν δράση μόνο για τι 10 ε, από αυτέ τι 300 και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δράσουν. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε τα κράτη θα μπορούν να εφαρμόσουν τα εθνικά τους μέτρα, θα πρέπει να στηρίζουν φυσικά αυτά τα μέτρα και με ποινικέ κυρώσει και με ε, διοικητικέ κυρώσεις εάν δεν υπάρχουν ε, κυρώσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και σε περιπτώσει όπου προβλέπονται ποινικέ κυρώσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα κράτη-μέλη δεν χρειαστεί να κάνουν τίποτα παραπάνω. Σα ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω με αυτόν τον τρόπο να απάντησα στις ερωτήσει των ευρωβουλευτών. Σα ευχαριστώ πολύ κυρία Κνούτσεν. Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος και αυτού του σημείου. Όπως είπε ήδη και ο κύριος Εποτάσιεβιτς, η παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης προβλέπεται για τις 19 Ιανουαρίου. Προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι στις 15 ε, Ιανουαρίου. Προτείνω λοιπόν να διακόψουμε για λίγα λεπτά και να συνεχίσουμε στις 10 ε, με την κοινή συνεδρίαση μαζί με τους συναδέλφου από τα Εθνικά Κοινοβούλια, όπου θα συζητήσουμε για την ε, ΣΥΠΟΛ και την Ευρωπόλ και την ανάκληση των αποφάσεων 371 και 681. Θα αρχίσουμε λοιπόν ξανά στις 10.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 Κυρίε Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας, αρχίσουμε, ας ε, συνεχίσουμε παρακαλώ την ε, συνεδρίαση. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξή μας είναι η συζήτηση για την Ευρωπόλ. Γνωρίζετε ότι η συνεργασία αυτή... Μήπως μπορείτε να καθίσετε παρακαλώ σιγά σιγά και να πάψει ο θόρυβος. Οι συζητήσεις παρακαλώ να διεξαχθούν έξω από την αίθουσα. Εκεί πίσω παρακαλώ. Ευχαριστώ. Το άρθρο 88 της Συνθήκης της Σαββόνας λέει καθαρά ότι η εποπτεία των δραστηριοτήτων της Ευρωπόλη διεξάγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Γι' αυτό η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών έχει προσκαλέσει όλα τα εθνικά κοινοβούλια να συμμετάσχουν στη σημερινή συζήτηση. Με μεγάλη χαρά λοιπόν καλωσορίζω σήμερα 7 συναδέλφους εθνικών βουλών, μεταξύ αυτών μάλιστα δύο πρόεδροι και ένας αντιπρόεδρος επιτροπών. Είμαι πολύ χαρούμενη που σας βλέπω σήμερα όλες και όλους εδώ και θα παρακαλέσω τους δικούς μου συναδέλφους ευρωβουλευτές να ενθαρρύνουν τους ε, δικούς τους εθνικούς βουλευτές να συμμετέχουν σε τέτοιες ε, συνεδριάσεις που εγώ βρίσκω πολύ σημαντικές. Υπάρχει ευρύ πεδίο συνεργασίας με ε, τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ελπίζω λοιπόν ότι η σημερινή συνεδρία δεν θα είναι η μοναδική, θα, θα ε, ακολουθήσουν και άλλες. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον εισηγητή και στους σκιώδεις εισηγητές και μετά θα δώσω το λόγο στους εθνικούς βουλευτές για τις δικές τους παρεμβάσεις. Όσοι εξημών επιθυμείτε να παρέμβετε, παρακαλείστε να ε, συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο και να το δώσετε στους ε, κριτήρες της αιθούσης οι οποίοι θα το παραδώσουν στη γραμματεία. Άρα λοιπόν παρακαλείστε να ε, προκαλέσετε το, την προσοχή των ε, κλητήρων για να έρθουν να λάβουν το έγγραφο. Και ε, θα αρχίσουμε με τον εισηγητή κύριο Διαστεμέρα. Διαστεμέρα, συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Α, πρώτα μου λόγια είναι για να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια για την παρουσία τους εδώ για το ζήτημα που θα συζητήσουμε σήμερα. Καλώς ήρθατε. Δεύτερον, θέλω να κάνω μια εισαγωγή σε σχέση με την νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχόλια που γνωρίζουν οι συνάδελφοι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά θα τα επαναλάβω έτσι ώστε να τα ακούσουν και οι συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια και να είναι πλήρω ενημερωμένοι. Εγώ ήμουν εισηγητή τη απόφαση του Συμβουλίου, εισηγητή ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με την απόφαση του Συμβουλίου. Η απόφαση του Συμβουλίου δεν ε, είναι συνεκτική με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτό ήταν μια μικρή παγίδα που μας έθεσε το Συμβούλιο, που θα θυμάται εκεί η Πρόεδρος, και τώρα διορθώνεται μέσω ενός κανονισμού, ο οποίος ε, πηγάζει από το πρόγραμμα της Στοκόλμης. Επομένως, ε, τώρα η συνθήκη της Λισαβόνας ενισχύει και αναγνωρίζει τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ποτέ δεν πρέπει να παραγωνίζονται. Η πρόταση κανονισμού της Ευρωπόλ αποτελείται από 14 κεφάλαια και 79 άρθρα. Εγώ ακολούθησα το εξή κριτήριο, θεματική διέρεση του κανονισμού σε πέντε σημεία. Το πρώτο σημείο έχει να κάνει με τις γενικές διατάξεις, τους ορισμούς και τους στόχους της Ευρωπόλ. Δεύτερον, έχουμε την συγχώνευση Ευρωπόλ σε πόλ όλοι εκτός από τους φιλελευθέρους είναι κατά της σε Ευρωπόλ σε Πολ, όλες οι ομάδες του Κοινοβουλίου. Εγώ ως εισηγητής είμαι ιδιαίτερα κατά. Λοιπόν, το τρίτο σημείο είναι η διακυβέρνηση. Κατόπιν έχουμε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο που θα το συζητήσουμε περαιτέρω στη συνέχεια. Και το τελευταίο, το πέμπτο, είναι πολύ σημαντικό θέμα για το Κοινοβούλιο και έχει να κάνει με την προστασία των δεδομένων εντός μιας υπηρεσίας ασφάλειας. Στις 18 Ιουνίου εγώ κατέθεσα την νομοθετική μου πρόταση μαζί με τις τροπολογίες. 125 τροπολογιε Σε τι συνίσταται διαγραφή κάθε αναφορά ψυχόνευση σε Ευρωπόλ, τροποποίηση διαγραφής για να δημιουργηθεί με εκτελεστική επιτροπή, δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Επίσης, ε, τροπολογίες για την ενίσχυση της προστασίας των δεδομένων της Ευρωπόλ, τροπολογίες ε, για να έχουμε ενίσχυση του ρόλου των εθνικών ε, ε, αρχών των εθνικών υπηρεσιών και τροπολογίες για να προωθήσω την εφαρμογή ενό αποτελεσματικού κοινοβουλευτικού ελέγχου. Στι 26 Σεπτεμβρίου έληξε η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών εδώ στο Κοινοβούλιο και πρέπει να σας ενημερώσω ότι οι συνάδελφοι παρουσίασαν 540 τροπολογίες και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτές με έναν απολυστευμένο τρόπο. Ο σκιώδης εισηγητής, ο κύριος Γιώσεφ Βάντεν Χόλφερ, 150, ε, η κυρία Αλφάνο 9, ο κύριος Κίρκοφ, 8, ο κύριος Ρούτα Βάρης 128 και η κυρία Χέρενς Κορνέλ 174. Από τις 540 τροπολογίες, 21 έχουν να κάνουν με στις γενικές διατάξεις, 32 με την απόρριψη της συγχώνευσης, 48 για τα καθήκοντα, 41 για τη διακυβέρνηση, 291 για την προστασία των δεδομένων. Αυτό μας δείχνει πόσο σημαντικά είναι για μας ε, τα θέματα αυτά της προστασίας των δεδομένων. 6 για την κατάργηση της εκτελεστικής επιτροπής, 10 για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο τρεις για τις οικονομικές διατάξεις και τέσσερις για τα παραρτήματα. Από τις 65 ε, για τα εκτιμώντα οι 10 αφορούν την απόρριψη της συγχώνευσης, 35 στην προστασία των δεδομένων, μία για την κατάργηση εκτελεστικής επιτροπής και υπόλοιπε 19 για τα υπόλοιπα θέματα. Η μέθοδο εργασίας που έχω ακολουθήσει έχει να κάνει με το να εξεύρω το δυνατότητα μεγαλύτερο αριθμό συμβιβαστικών τροπολογιών. Γι' αυτό ήδη συναντήθηκα δύο φορές με τους σκιώδεις συζητητές και χάρη σε αυτό πρότεινα 22 συμβιβασμούς. Ο πρώτος αναφέρεται στις 42 τροπολογίες σχετικά με την κατάργηση όλων όσων έχουν να κάνουν με τη συγχώνευση σε πόλευρο πόλη. Δεύτερον, ένας μόνος συμβασμός για 7 τροπολογίες που έχουν να κάνουν με την κατάργηση της δημιουργίας μιας εκτελεστικής επιτροπής, που εμείς δεν θεωρούμε απαραίτητη. 20 υπόλοιποι συμβιβασμοί έχουν να κάνουν με τις γενικές διατάξεις, τους ορισμούς, τους στόχους της Ευρωπόλ και τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω τους κοιόδης εισηγητές ε, για την τόσο πολύπλοκη και επαγγελματική δουλειά τους. Και όπως ε, σας εξήγησα θα συνεχίσω να καλώ συνεδριάσεις ε, για να σημειώσουμε πρόοδο στην ανάπτυξη της νομοθετικής πρότασης σαν Η επόμενη συνάντηση είναι στις 4 Δεκεμβρίου και θα ασχοληθούμε με το θέμα του κοινοβουλευτικού έγχου για να εξετάσουμε εκεί όλες τις τροπολογίες που υπάρχουν σχετικά με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και τέλος, νομίζω ότι θα έχουμε πολλές συναντήσεις για να συζητήσουμε την ουσία του θέματος και το θέμα της προστασίας των δεδομένων εντός μιας υπηρεσίας ασφαλείας. Έχοντας ε, υπόψη την παρουσία των συναδέλφων από τα Εθνικά Κοινοβούλια, θα ήθελα να προσδώσω ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα του κοινοβουλευτικού ελέγχου προκειμένου να προσαρμόσουμε την Ευρωπόλη στις απαιτήσεις της συνθήκης της Λισαβόνας, ο κανονισμός εγγυάται μέσω των δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες Ευρωπόλη να υπόκειται στο δημοκρατικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Αυτός ο έλεγχος αναφέρεται συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 9 της πρότασης κανονισμού. Αν έχουμε και πολυάριθμες αναφορές ε, σε αυτόν τον έλεγχο, σε όλο το διατακτικό. Ο μηχανισμός ελέγχου ήταν δραστηριοτήτων της Ευρωπόλα από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων και έχω κάνει κάποιες τροπολογίες, προτείνω να γίνει μέσα από μια συγκεκριμένη δομή που θα στελεχώνεται από την αρμόδια επιτροπή, την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ δηλαδή, και θα συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής, της Εσωτερικής Επιτροπής Δικαιοσύνης ε, από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αυτός ο έλεγχος πάντοτε θα γίνεται εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα καλούνται οι συνεδριάσεις από τον πρόεδρο της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και θα συμπροεδρεύει και ένας εκπρόσωπος των Εθνικών Κοινοβουλίων που θα λαμβάνει την Προεδρία Εκπεριτροπής στο Συμβούλιο. Τι θέλουμε να κάνουμε τώρα λοιπόν με αυτή την ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου. Θα παρουσιάσουμε εκεί το, θα παρουσιαζόταν εκεί η έκθεση δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ, το ετήσιο και πολιετές ε, πρόγραμμα της Ευρωπόλ. Όταν λέω να παρουσιάσετε, θα παρουσιάσετε, θα συζητείτε κιόλα. Η ε, έκθεση του Ευρωπαίου την Προστασία των Δεδομένων, η έκθεση αξιολόγηση που κάνει η Κομισιόν κάθε πέντε χρόνια για την αποτελεσματικότητα της Ευρωπόλ. Επίσης, αυτή η δομή ελέγχου θα μπορούσε να καλέσει τον υποψήφιο εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπόλ για να υπάρχει μια κρόση εδώ και να κάνει μια δήλωση ο άνθρωπος αυτός, αλλά και να ενημερώσει σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του. Επίσης, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο εκτελεστικός διευθυντής, ο Ευρωπαϊκός Επόπτης των Ευρωπαϊκών Συνδεδομένων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμμετέχουν σε αυτές τις συζητήσεις. Επίσης, τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Εθνικό Κοινοβούλιο θα ενημερώνονται σχετικά με την αξιολόγηση των απειλών και των κινδύνων, τις στρατηγικέ αναλύσεις και τις γενικές εκθέσεις που σχετίζονται με τους στόχους της ε, Ευρωπόλ και τα αποτελέσματα των μελετών και των αξιολογήσεων που θα έχουν αναλυφθεί. Και θα ολοκληρώσω εδώ αλλά θα ήθελα να αναφέρω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να λειτουργεί και ως αρμόδιο όργανο δημοσιονομικού ελέγχου και θα πρέπει να λαμβάνει την, και να αξιολογεί την έκθεση για την δημοσιονομική διαχείριση και επίσης ε, είτε θα εγκρίνουμε είτε θα απορρίπτουμε τη διαχείριση του εκτελεστικού διευθυντή και διαχείριση του οργανισμού. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Τώρα, προς ενημέρωσή σας και προς ενημέρωση των συναδέλφων ε, που βρίσκονται από τα Εθνικά Κοινοβούλια, θα καλέσω τον εκπρόσωπο της Λιθουανικής Προεδρίας να ε, παρέμβει πρώτος. Πρωτού δώσω το λόγο στους ευρωβουλευτές και στα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων. Θα έχει ο καθένα από εσά τρία λεπτά χρόνο ομιλία, έτσι ώστε να ε, διεξάγουμε την συζήτηση στο χρόνο που έχει προβλεφθεί. Τώρα θα, δώσω, θα δώσω το λόγο στην κυρία Βικτόρια Μιξίτα, που είναι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να απαντήσει στον εισηγητή. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι όντω πολύ σύντομη. Σε αυτό το στάδιο θα περιοριστώ στα ακόλουθα σχόλια. Καταρχάς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι ο αριθμός και η σημασία που έχουν οι τροπολογίες που έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα από τον εισηγητή και από τα άλλα μέλη της Επιτροπής είναι μια μαρτυρία του ενδιαφέροντος και της δέσμευσης της Επιτροπής αυτής για να διαμορφώσει την νομοθεσία για κάτι τόσο σημαντικό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό όργανο συνεργασίας στον ε, τομέα της επιβολής του νόμου, της Ευρωπόλη δηλαδή. Όπως ε, τόνισε ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες της πρότασης αυτής πράγματι σχετίζεται με τον ε, στόχο του να γίνει η Ευρωπόλη ένα και περισσότερο υπόλογη στο Ευρωκοινοβούλιο, στα Εθνικά Κοινοβούλια και στους Ευρωπαίους πολίτες. Επίσης εδώ να σημειώσουμε ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ για το ότι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια έχει ε, προσελκύσει τόσο ενδιαφέρον. Τώρα, όσον αφορά τις υπόλοιπες ε, πτυχές αυτής της πολύ σημαντικής πρότασης, να πω ότι θα ακούσουμε με μεγάλη προσοχή την ε, συζήτηση που θα ακολουθήσει. Και χαιρόμαστε πολύ και για τους ε, ενδεχόμενους συμβιβασμούς που θα υποβάλει ο κύριος Δίας Δεμέρα σε αυτή την Επιτροπή μετά από την συνεργασία του με τους συναδέλφους και τους κοιόδες εισηγητές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα ήθελα να καλέσω την κυρία Πολιάκα από την Λιθουανική Προεδρία να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και εγώ θα είμαι σύντομη σε αυτό το στάδιο. Θα ήθελα απλά να επιβεβαιώσω ότι το Συμβούλιο έχει ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα όσον αφορά αυτό το σχέδιο κανονισμού και έχουμε καταφέρει να έχουμε αρκετή πρόοδο στην άρθρο προς άρθρο ανάλυση της πρότασης αυτής. Και για μας ισχύει η ίδια αρχή, η ίδια προσέγγιση, ακολουθούμε την ίδια γραμμή, αλλά προσπαθούμε να βρούμε όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία συμβιβασμού στο Συμβούλιο, αλλά και σε συνεργασία με την επόμενη Προεδρία θα είμαστε σε θέση να εισέλθουμε σε επίσημο διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζουμε να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα αρχίσει η συζήτηση. Αρχίζουμε με τους κοιόδες εισηγητές. Κύριε Βάιντεν Χόλτσαρ, έχετε τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κανονισμός της Ευρωπόλ είναι μια πάρα πολύ σημαντική νομική πράξη που δυστυχώς ε, έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αφορά την ασφάλεια και την ασφάλεια δικαίου και υπάρχουν πολύ σημαντικές ε, πτυχές που πρέπει να είναι προϋπόθεση για την ασφάλεια. Ε, η λισαβονοποίηση της Ευρωπόλ με αυτόν τον κανονισμό δεν είναι ε, σκοπός του κανονισμού αυτού. Ο σκοπός και στόχος είναι να γίνει η Ευρωπόλη πιο αποδοτική στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας ε, και για την διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων. Έχει βρεθεί μία μέθοδος εργασίας η οποία είναι αρκετά ε, γρήγορη. Έχουμε αποφασίσει, έχουμε συμφωνήσει για αρκετούς συμβιβασμούς σε πολλούς τομείς. Ορισμένα σημεία θα ήθελα τώρα να αναφέρω για εμένα και για την ε, κοινοβουλευτική μου ομάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα σαφή διαχωρισμός σε Ευρωπόλ και σε Πολ. Δεν θεωρούμε πως είναι σωστό αυτές οι δύο υπηρεσίες να συγχωνευτούν. Πιστεύουμε πως ε, έχουν ε, διαφορετικά χαρακτηριστικά έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες και είναι πάρα πολύ επίσης σημαντικός ο κοινοβουλευτικό έλεγχος και η πρόταση του ε, εισηγητή να συσταθεί μία επιτροπή ελέγχου από την δική μας επιτροπή είναι κάτι που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και πιστεύω πως ε, συνάδει και με το πνεύμα της συνθήκης της Λισαβόνας. Ε, πιστεύω πως θα καταφέρουμε να βρούμε έναν τρόπο λειτουργίας αποτελεσματικό, θα καταφέρουμε να συστήσουμε μια επιτροπή η οποία θα μπορέσει να ε, δρομολογήσει τον κανονισμό σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν πάρα πολλές ε, διοικητικές ε, δυνατότητες που μπορούμε να εγκρίνουμε. Είναι πολύ σημαντικό το Κοινοβούλιο να έχει σημαντικό ρόλο επόπτη και παρατηρητή. Επίσης, ε, όσον αφορά την Εκτελεστική Επιτροπή, εγώ προτείνω επίσης να διαγραφεί, διότι πιστεύω πως δεν επιφέρει καμία βελτίωση ε, των δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ. Ε, πολύ σημαντικές επίσης είναι και οι διατάξεις για την προστασία των δεδομένων. Έχουμε συζητήσει εκτενώς με τον εισηγητή για το θέμα αυτό. Είναι πολύ σημαντικές όπως είπα ε, και πρέπει να ε, συνδεθούν οι διατάξεις αυτές και με την αντίστοιχη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. ιδιαίτερα στο σημείο, στο θέμα της ανταλλαγής δεδομένων με τις ε, εθνικές κυβερνήσεις και με ιδιωτικού ε, φορείς. Εμείς καλούμε για μία αξιολόγηση και έλεγχο. διότι δεν είμαστε σίγουροι εάν εφαρμόζονται τα ευρωπαϊκά πρότυπα στην ε, ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα σε ιδιωτικούς, ε, από ιδιωτικού φορεί. Είναι επίση πολύ σημαντικό να συζητήσουμε εκτενώ ε, για την προστασία δεδομένων και για το ρόλο του επόπτη προστασίας δεδομένων. Είναι μια θέση πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει να είναι ανεξάρτητη και είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπόλ να βρίσκεται στον συντονιστικό ρόλο. Εύχομαι τέλος να υπάρξει το κατάλληλο ενδιαφέρον και από τα εθνικά κοινοβούλια, ώστε να υπάρξει και η βέλτιστη συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφα. Θα ήθελα να πω στους συναδέλφους ότι εάν καταφέρουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα θα καταφέρουμε να έχουμε και ένα δεύτερο κύκλο ε, συζήτησης. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθώ να σας περιορίσω Κύριε Κέρκοπ, έχετε τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι ε, εγκρίνω και συμφωνώ στα πάντα όσον αφορά την Ευρωπολή. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική υπηρεσία και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την συνεργασία της ε, δικής μου χώρας με το έργο της Ευρωπόλ. να στηρίξουμε επίσης τον ελέγχιστο, την ελέγχιστη κατανομή πόρων. Η Ευρωπόλ έχει αναλάβει παραπάνω καθήκοντα την ε, Συμφωνία για τα Δεδομένα των Επιβατών και άλλες συμφωνίες οι οποίες επιφέρουν περισσότερο ε, φόρτο εργασίας. Ωστόσο, θα ήθελα να σχολιάσω κυρίως το θέμα του ελέγχου Έχω επιχειρηματολογήσει και στο παρελθόν ενώπιον του Κοινοβουλίου για το ότι δεν θέλω να πολιτικοποιηθεί η Ευρωπόλη. Δεν θέλω να δω μια Ευρωπόλη η οποία θα υπόκειται είτε σε ευρωπαϊκό, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε σε κάποιον ευρύτερο φορέα. Δεν θέλω να δω ε, κανόνες που θα είναι περιοριστικοί όσον αφορά τον έλεγχο, κανόνες οι οποίοι θα κάνουν πιο δύσκολο το έργο της Ευρωπόλη από ό,τι στο παρελθόν. Έχω παρευρεθεί σε συνέδρια που συμμετείχαν και τα Εθνικά Κοινοβούλια και πιστεύω πως ε, δεν ε, αναφέρομαι μόνο στην άποψη του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και στις ε, απόψεις άλλων κρατών. Πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη να, να μοιράζονται τις αρμοδιότητες του ελέγχου και να είμαστε σαφείς για το τι αρμοδιότητες θα έχει ο καθένας προτού προχωρήσουμε σε μία πρόταση. Πρέπει να δείξουμε μεγάλη προσοχή. Και να προσθέσω στο σημείο αυτό ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί να μην περιορίσουμε τις αρμοδιότητες της Ευρωπόλου διότι προκύπτουν νέες προκλήσεις ε, συνεχώς και δεν θα ήθελα να βρεθούμε σε μια ε, κατάσταση όπου η Ευρωπόλη δεν θα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει, όπου θα παρατηρούνται καθυστερήσεις που δεν θα είναι αναγκαίες, όλα αυτά εξαιτία του ελέγχου. Πιστεύω ότι οτιδήποτε κάνει πιο πολιτικοποιημένη την Ευρωπόλ θα με δυσαρεστήσει πάρα πολύ. Θα ήθελα τα ζητήματα που θα συζητηθούν να έχουν περισσότερο να κάνουν με την εύρυθμη λειτουργία της Ευρωπόλ. Εντάξει, μπορώ να δεχτώ ότι είναι επιθυμητή έτσι κάποια μορφή ελέγχου, αλλά να πιστήσω την προσοχή στην, στο μέτρο. Ευχαριστώ πολύ κυρία, κυρία Κέρκοπ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι ευχαριστήσεις μου πηγαίνουν πρώτα στον εισηγητή. Η βάση που μας έδωσε για τη συζήτηση μας ικανοποιεί. Γνωρίζουμε ότι η Ευρωπόλ, η έκθεση για την Ευρωπόλ δηλαδή είναι από τις πιο σημαντικές που συζητούμε εδώ, σε ολόκληρη την κοινοβουλευτική θητεία. Γνωρίζουμε και πόσο επικρίνεται η Ευρωπόλ, ιδίω για την έλλειψη διαφάνεια, που είναι αυτό που μα ανισχύει περισσότερο. Και στο κάτω τη γραφή δεν υπάρχει και δυνατότητα ελέγχου. Εκεί εντοπίζεται η κριτική μα. Και το βλέπουμε όταν έρχεται ο κ. Wainwright εδώ και μα απευθύνει το λόγο. Θέλουμε λοιπόν να αποσαφινιστούν τα θέματα αυτά. Τώρα για τα επιμέρους. Εμείς ως Ενωτική Αριστερά ενδιαφερόμαστε αφενός για το πεδίο εφαρμογής. Δηλαδή, ποιο θα είναι αυτό. Ωραία, ο οργανωμένο έγκλημα σύμφωνη. Βαρύ οργανωμένο έγκλημα επίσης σύμφωνη. Αλλά πόσο ευρύ είναι το πεδίο αυτό εφαρμογής. Γι αυτό, αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό. Αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει με άνεση χρόνου και να μην μείνει μονάχα στην Ευρωπόλη. Για την ΕΑΑ τώρα, για την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία, συμφωνούμε. Θεωρούμε ότι δεν έχει νόημα να συγχωνευτεί και απορρίπτουμε αυτά που προωθούν με τέτοια ένταση Συμβούλιο και Κομισιόν. Τρίτο, κοινοβουλευτικός έλεγχος. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι χρειάζεται ένα ελεγκτικό όργανο με μια συγκεκριμένη σύνθεση, περιορισμένη σύνθεση και ιδίω να κατοχυρωθεί ως ελεγκτικό όργανο, δηλαδή θα μπορούσαν ίσως να είναι και ένα ή μόνο δύο μέλη από μια πολιτική ομάδα, αλλά με πλήρη δικαιώματα, δηλαδή ξεκάθαρα δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα εξέταση των εγγράφων όχι απλά η υποβολή ερωτήσεων στην Ευρωπόλ, η οποία θα απαντήσει όπως θέλει, αλλά να τους δοθεί η δυνατότητα πραγματικά να απαιτήσουν και να λάβουν αληθείς απαντήσεις. Διότι εν τέλει πρόκειται για το δικαίωμα πληροφόρησης του ίδιου του Κοινοβουλίου. Βεβαίω είναι σημαντικό να συμμετάσχουν και τα εθνικά κοινοβούλια, σωστό, όμως δεν μπορούν να αποφασίζουν. Μόνο συμβουλευτικά. Να συντονιστεί ο διάλογος μεταξύ των ε, κοινοβουλίων, ναι, σωστό. Να σκεφτούμε λίγο και τη συζήτηση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης που υπάρχει εδώ εγγράφος και να αντιδράσουμε. Όπως είπα, να λάβουμε όσο χρόνο χρειάζεται. Χαίρομαι που ο εισηγητής στάσεται υπέρ του κοινοβουλευτικού ελέγχου και εμείς θα υποστηρίξουμε κάθε κίνηση προς την κατεύθυνση αυτή. Τέλος, προστασία δεδομένων. Εμείς βεβαίως θα απαιτήσουμε να είναι εξασφαλισμένη η προστασία αυτή. Όχι εκτελεστική επιτροπή, σε αυτό συμφωνούμε. Υπάρχουν πολλά σημεία συμφωνίας. Εμείς πάντως θα επιμείνουμε και θα εμείνουμε πολύ στον έλεγχο. Βεβαίω, αυτά θα τα πούμε και στις ε, συνεδριάσεις των συντονιστών και σκιωδών μάλλον. Ευχαριστώ. Έρχομαι τώρα στον μεικτό κατάλογο αγοριτών και διαβάζω τα ονόματα. Lord Hanna for the UK, Mr. Cengar Zalan for Hungary, Madame Mathieu, Mr. Latskovskis from Latvia, Madame Caramondi from France and myself. Is there anybody else who... Και εγώ ίδια. Άλλος κανείς επιθυμεί να παρέμβει? Ο κύριος Μισελ. Από τις Εθνικές Βουλές. Άλλος κανείς? Εφόσον επιθυμείτε, παρακαλώ, κάνετε νόημα στους κλητήρες ή και στη γραμματεία. Θα αρχίσουμε λοιπόν με τον ε, Μιλόρδο Χάνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις αφού πρώτα καταστήσω σαφές ότι μιλώ για τα άρθρα μόνο 53 και 54 του κανονισμού. Και τροπολογίες 626-634. Διότι βέβαια η Βρετανική κυβέρνηση αρμόζει να μιλήσει για τα βασικότερα θέματα και όχι εγώ, όσα δηλαδή θα συζητηθούν στο Συμβούλιο. Και εμείς έχουμε υποβάλει τις απόψεις μας στη Βρετανική κυβέρνηση σχετικά. Δεν νομίζω όμως ότι είναι σκόπιμο ε, για μένα να επεκταθώ σε αυτά. Δεύτερο, είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για τον προσεκτικό και πλήρη τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και εσείς κυρία Πρόεδρε περιλάβατε τις Εθνικές Βουλές στα θέματα των ρυθμίσεων του κοινοβουλευτικού ελέγχου επί της Ευρωπόλ. Νομίζω ότι είναι καινοτόμο ο τρόπος με τον οποίο εσείς αναγνωρίζετε ότι βρισκόμαστε σε χώρο μεικτών ε, κοινών αρμοδιοτήτων και ότι τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια δηλαδή έχουν γνήσιο καθεστώς εν προκειμένου. Και οι ρυθμίσεις θα είναι στέρεες μόνον εφόσον συνδυαστεί η εργασία των Εθνικών Βουλών με της Ευρωπαϊκής. Σας ευχαριστώ λοιπόν που αναγνωρίζετε το γεγονός αυτό. Ε, μάλιστα νομίζω η τρίτη συνεδρία στη σημερινή και τη θεωρώ πραγματικά πολύτιμη. Οι απόψεις της Βουλής των Λόρδων καταστρώθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου φέτος όταν ο Λόρδος Μπόζελ, ο πρόεδρος της ε, συνολικής μας Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων έστειλε επιστολή στον εισηγητή σας που περιλαμβάνει πλήρως τις απόψεις μας και θεωρώ ότι σας είναι οικίες. Εμένουμε στις απόψεις αυτές. Θεωρούμε ότι ο μηχανισμός εποπτείας θα πρέπει να είναι ελαφρός, light, να αποφύγει την δημιουργία νέων οργάνων και να βασιστεί στις υφιστάμενες συνεδριάσεις μεταξύ της Επιτροπής, ε, ε, μεταξύ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και των συναρμόδιων επιτροπών των Εθνικών Κοινοβουλίων, που νομίζω ότι το σύστημα αυτό λειτουργεί. Και ωστόσο εξακολουθεί και δεν είναι βαρύ. Πιστεύουμε ακόμη, και αυτό είναι το δεύτερο σημαντικό θέμα, ότι η κοινοβουλευτική εποπτεία θα πρέπει να αποφύγει η παρέμβαση στο επιχειρησιακό έργο της Ευρωπόλ. Πώς λοιπόν συναρμόζονται οι τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, αυτό μας ρωτάτε σήμερα, με τους στόχους που προανέφερα. Μου φαίνεται ότι η προτινόμενη Επιτροπή Κοινοβουλευτικού Ελέγχου καλά τα καταφέρνει. Έχω βέβαια κάποια σχόλια σχετικά. Ένα σημείο κριτική είναι ότι ίσως, ίσως είναι κατανοητό βέβαια, ότι ο εισηγητή έχει μεταφέρει κάπως την διαχείριση της Επιτροπής αυτής, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και απομακρύνοντα την από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και νομίζω ότι και η Γαλλική Εθνοσυνέλευση και η Ιρλανδική Βουλή έθεσαν τα θέματα αυτά και εγώ συμφωνώ με τι απόψει του. Είναι σημαντικό να θυμηθεί κανείς ότι έχουμε μπροστά μας δραστηριότητες, πολλές από τις οποίες παραμένουν ξεκάθαρα μέσα στα πλαίσια αρμοδιοτήτων των χωρών μελών και που πιθανότατα έτσι θα παραμείνουν και στο προσεχές μέλλον. Άρα οι διαδικασίες της Επιτροπής αυτής θα πρέπει να είναι αλλά και να φαίνονται καθαρά ότι είναι εξισορροπημένες. Επίσης είναι σημαντικό να θυμηθεί κανείς, όπως άλλωστε το είπε προς το τέλος της παρεμβάσεώς του και ο ίδιος ο εισηγητής και νομίζω ότι πολύ σωστά έπραξε, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη διαθέτει ένα προνόμιο μέσω της ε, δημοσιονομικής διαδικασίας, του προπολογισμού, στην οποία δεν έχουν καμία πρόσβαση οι Εθνικές Βουλές. Και έτσι θα συνεχίσει να είναι. Νομίζω οι νέες ιδέες που προτείνονται τώρα για την εποπτεία θα πρέπει να είναι πολύ πιο εξισορροπημένες από ό,τι τώρα στο σχέδιο. Δεύτερο, ερχόμαστε στην προτινόμενη μονάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου που είναι κάτι διαφορετικό. Δεν θέλω να σας κρύψω ότι έχω σημαντικότατες επιφυλάξεις ακόμα και για την ίδια την ύπαρξη της μονάδας αυτής και όχι καν για τις αρμοδιότητές της που περιλαμβάνονται στις τροπολογίες και που όπως είναι οι τροπολογίες ενισχύουν τις επιφυλάξεις μου διότι η προτινόμενη εντολή θα δώσει στη μονάδα αυτή αρμοδιότητες που ούτε καν διανοούνται να ασκήσουν τα εθνικά κοινοβούλια απέναντι στις ανεξάρτητες αστυνομικές αρχές. Προσοχή λοιπόν, οποιαδήποτε κίνηση προς την κατεύθυνση αυτή θα μας βρει αντίθετους. Η Ευρωπόλ μου φαίνεται ότι είναι σημαντικό, πολύτιμο εργαλείο, οργανισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται την κοινοβουλευτική εποπτεία και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τα εθνικά. Δεν το αμφισβητώ αυτό αλλά χρειάζεται επιχειρησιακή αυτονομία, όπως ε, διαθέτουν και οι εθνικές αστυνομικές αρχές. Ελπίζω να καταφέρετε να τετραγωνίσετε λοιπόν τον κύκλο αυτό, έτσι ώστε να ωφεληθούμε όλοι. Σας ευχαριστώ. Καθώς ε, πρόκειται για μια ειδική συνεδρίαση και δεν θέλω να είμαι αγενής ε, στους προσκεκλημένους μας, δεν σας διέκοψα, αλλά θα ήθελα να σας απευθύνω έκκληση, να σεβαστείτε τα τρία λεπτά και αν υπάρχει χρόνος μπορείτε να επανέλθετε. Να δευτερολογήσετε, δεν θα είναι πρόβλημα αυτό αλλά σας παρακαλώ προσπαθήσουμε να σεβαστούμε το χρόνο. Από την Ουγγαρία, και συγγνώμη αν δεν προφέρω σωστά το όνομά σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ευχαριστώ εξάλλου και για την πρόσκληση που απίφθινε η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και είναι τιμή για μας να παρευρισκόμαστε. Η Ευρωπόλ είναι ευρωπαϊκός οργανισμός ο οποίος λειτουργεί ορθά. Σύμφωνη, ε, Σύμφωνα με την συνθήκη της Λισαβόνας βέβαια απαιτούνται ορισμένες τροποποίησεις. Νομίζω ότι η πρόταση της Κομισιόν ωστόσο υπερβαίνει την ανάγκη αυτή. Θα τονίσω ορισμένα πράγματα. Πρώτα, εκπαίδευση και κατάρτιση, και διαρκής κατάρτιση. Η Ουγγαρία είναι υπέρ της ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας. Δεν είμαστε υπέρ της συγχώνευσης. Το επιχείρημα το οποίο ε, προβάλλεται είναι το δημοσιονομικό, δηλαδή για λόγους οικονομίας. Εγώ θεωρώ ότι δεν ε, αρκεί το επιχείρημα αυτό. Η κατάρτιση ανήκει στην ε, Ευρωπαϊκή Αστυνομική Αστυνομία. Οποιαδήποτε συγχώνευση ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανεξαρτησία των οργανισμών αυτών. Οι δύο οργανισμοί διαθέτουν, μάλλον έχουν διαφορετικές λειτουργίες. Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάρτιση βλέπουμε και επιχειρήματα τα οποία οδηγούν να θεωρήσουμε ότι είναι καλύτερο να παραμείνουν ξεχωριστοί οι δύο οργανισμοί. Επίσης, εφόσον συγχωνευτούν οι δύο οργανισμοί, θα ζημιωθεί η διαφάνεια. Υπενθυμίζω την συνάντηση στις 8 Δεκάτου των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι ζήτησαν η, Ευρωπόλ, ε, συγγνώμη, η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία να λάβει έδρα στην Βουδαπέστη. Ελπίζω ότι αυτό θα επιτευχθεί. Σε ό,τι αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, να μην λησμονούμε την απόφαση της 11 Απριλίου 2011 η διακοινοβουλευτική συνεργασία θα συνεχιστεί με συμμετοχή όλων των μερών. Ε, εγώ θεωρώ ότι όλοι τάχθηκαν υπέρ τότε της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος της Ευρωπόλ διεξάγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τα Εθνικά. Διότι το άρθρο 88 για τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνθήκης δηλαδή, λέει ότι κοινοβουλευτικός έλεγχος, ο κοινοβουλευτικό έλεγχος δεν ασκείται ορθά για την ώρα. Γι' αυτό θα καταστεί απαραίτητο να ιδρυθεί διακοινοβουλευτικό όργανο με συμμετοχή ευρωβουλευτών και, βουλών των, και ε, βουλευτών των Εθνικών Βουλών. Και οι πρόεδροι των Βουλών θα πρέπει να ορίσουν την σύνθεσή του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στην κυρία Ματιά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Είναι πάντοτε μεγάλη ικανοποίηση να συνεργαζόμαστε από κοινού ενός ε, επί ενό νομοθετήματο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλω να ευχαριστήσω και τον συγητή και τους κοιόδε εισηγητές. Ο κύριος Βέντενχόλσον μα είπε ότι υπήρχε καθυστέρηση, ναι, είναι αλήθεια γιατί τώρα καθυστέρησε αυτή η πρόταση της Κομισιόν, γιατί στην αρχή, και το γνωρίζετε καλά, είχαμε δύο προτάσεις. Την πρόταση περί σε ΣΕΠΟΛ, της αναθεώρησης της ε, νομικής βάσης για τη ΣΕΠΟΛ και για τη λισαβονοποίηση Τη Ευρωπόλ και κατόπιν άλλαξε γνώμη η Κομισιόν και μα είπε τελικά θα συγχωνεύσουμε την ε, ΣΕΠΟΛ και την Ευρωπόλ. Το Κοινοβούλιο όρισε τον εισηγητή για τη ΣΕΠΟΛ, ε, οι πολιτικές ομάδες διόρισαν τους κοιόδης εισηγητές ε, και τελικά και τον εισηγητή για την Ευρωπόλ και τελικά βρεθήκαμε εν ώψη εκπλήξεως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μας παρουσίασε την πρόταση συγχώνευσης. Ο εισηγητής και σκιώδης εισηγητής της ΕΠΟΛ δεν είχαν πλέον πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αστυνομική Ακαδημία και ακούσαμε ότι είπαν οι συνάδελφοι του Ελληνικού Κοινοβούλου ίσως θα υπάρχει πρόταση από το Συμβούλιο και ίσως να μπορέσουμε να εργαστούμε επί της πρότασης αυτής και αυτό θα είναι καλό γιατί εμείς πράγματι είμαστε αντίθετοι στη συγχώνευση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία γιατί η αστυνομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται μια ανεξάρτητη και πραγματική κατάρτιση και η ΣΕΠΟΛ ε, πρέπει να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά της που την κάνει πολύ καλά. Πρόκειται μια πολύ καλή υπηρεσία για ένα πολύ καλό οργανισμό και η Ευρωπόλ από την άλλη είναι μια υπηρεσία που έχει μια πολύ σημαντική αποστολή και φυσικά πρόσφατα η Κομισιόν ε, της ανέθεσε και την καταπολέμηση του εγκλήματος στο κυβερνοχώρο και της καταπολέμησης ε, του εις όπλων, του της παράνομης διακίνησης όπλων. Νομίζω λοιπόν ότι οι δύο αυτοί οι οργανισμοί θα πρέπει να παραμείνουν ανεξάρτητοι για να μπορούν να εκπληρώνουν κατάλληλα τα καθηκοντά τους. Έτσι λοιπόν, ε, οι προτάσεις του εισηγητή και των σκεδών είναι πολύ σημαντικές, νομίζω, πως ε, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στον τρόπο με τον οποίο εργάζεται η Ευρωπόλ και θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στην Ευρωπόλ να συνεχίζει να εργάζεται σωστά χωρίς να θέτουμε εμπόδια στην ορθή της λειτουργία. Θα πρέπει ε, να δούμε βέβαια και το θέμα της επεξεργασίας των δεδομένων. Να προσπαθήσουμε να συζητήσουμε με τον Οργανισμό Προστασίας των Δεδομένων έτσι ώστε να εκπονήσουμε την ε, κατάλληλη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων χωρίς βέβαια όπως σας είπα να εμποδίσουμε το έργο της Ευρωπόλ. Και σε ό,τι αφορά την καλή διακυβέρνηση νομίζω ότι κανείς δεν παραπονιέται γι' αυτό σήμερα. Ναι, μεν, θα πρέπει να τροποποιήσουμε τον τρόπο που γίνεται ο κοινοβουλευτικό έλεγχο, αλλά νομίζω ε, τα όσα είπε ο εισηγητή σήμερα είναι λογικά, είναι λογικέ οι προτάσει αυτέ και δεν θα ήθελα να έχουμε ένα πιο βαρύ έλεγχο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις διεθνείς συμφωνίες, θα πρέπει να δούμε και με ποιους όρους θα συνάπτονται συμφωνίες στο μέλλον, αλλά ο χαρακτήρας δηλαδή το να έχει αναδρομική ισχύ, ε, μου φαίνεται δύσκολο. και νομίζω ότι θα είναι μακρύς διαπραγματεύσεις και θα μπορούσαν να κρατήσουν πολύ χρόνο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Λατσκόσκης από την Λετωνία. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη για κοινοβουλευτικό έλεγχο, αλλά ο έλεγχος θα πρέπει να οργανωθεί εντός των φυστάμενων κοινοβουλευτικών δομών. Δεν βλέπουμε λοιπόν να υπάρχει καμία ανάγκη για τη δημιουργία μιας νέας κοινοβουλευτικής μονάδας. Πιστεύουμε ότι η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Κοινοβουλίου σας θα μπορούσε να διοργανώσει κοινέ συνεδριάσεις με την Ευρωπόλ και με τις αντίστοιχες επιτροπές των Εθνικών Κοινοβουλίων και ταυτόχρονα οι επικεφαλής οι πρόεδροι των Επιτροπών Εσωτερικών Υποθέσεων από τα Εθνικά Κοινοβουλία θα μπορούσαν να οργανώνουν συχνές συναντήσεις με την Ευρωπόλη. Υπάρχουν και άλλες δυνατότητες που προτάθηκαν από τους συναδέλφους από τα κράτη-μέλη και νομίζω ότι αυτές οι προτάσεις θα πρέπει επίσης να εξεταστούν από την Επιτροπή σας. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαστε πολύ σύντομος, κυρία Καραμανλή από τη Γαλλία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση να συμμετέχουν οι εθνικοί δουλευτές στη συνεργασία με το, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό το σχέδιο κανονισμού είναι σημαντικό. Θα αναφερθώ σε τρία σημεία. Το πρώτο αφορά τη συγχώνευση των δύο υπηρεσιών και εμεί δεν θεωρούμε ότι είναι σκόπιμη η συγχώνευση για τους λόγους που αναφέρθηκαν από τους υπόλοιπους συναδέλφους. Τώρα για τις υπόλοιπες διατάξεις, για τη διαβίβαση των πληροφοριών, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι οι διατάξεις που προβλέπονται σήμερα κατά την άποψή μας δεν επαρκούν και η έγκριση ενός κράτους μέλους ε, δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Θα πρέπει λοιπόν ρητά να δίνεται κάθε φορά αυτή η έγκριση για τη διαβίβαση των πληροφοριών. σε ό,τι αφορά το θέμα της διακυβέρνησης, αφού διαβάσαμε το σχέδιο έκθεσης ε, του κυρίου Ντία Δεμέρα, ο οποίος έχει προβεί σε μια σειρά τροποποιήσεων, θεωρούμε ότι θα μπορούσαν να εξελιχθούν κάποια σημεία. Δηλαδή, ο ε, υποψήφιος που θα έχει επιλεχθεί για τον εκτελεστικό διευθυντή θα κληθεί για μια ακρόαση. Εμείς πιστεύουμε ότι ίσως θα ήταν καλύτερο να προβλέψουμε μια γνωμοδότηση της μονάδας κοινοβουλευτικού ελέγχου ε, πριν αποφασιστεί ε, η επέκταση της θητείας τους και επίσης το ίδιο να ισχύει πριν ε, το Διοικητικό Συμβούλιο πάυσει τον εκτελεστικό διευθυντή. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Εδώ διαβιβάσαμε το ψήφισμα που εθετήθηκε χθε από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και θα συζητηθεί από την Επιτροπή Νομοθεσίας όπου συμμετέχω και εγώ και εμείς η Γήτρια. Είμαστε υπέρ του να δημιουργηθεί μια μεικτή επιτροπή που θα συμμετέχουν βουλευτέ και από τα Εθνικά Κοινοβούλια και από τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια. Αυτή η μεικτή επιτροπή θα έπρεπε επίση ε, να ε, αποτελείται και από μέλη τη Επιτροπή ΛΥΜΠΕ αλλά και από εθνικού βουλευτέ που είναι αρμόδιοι για το θέμα τη εσωτερική ασφάλεια και θα πρέπει να συμμετέχουν ε, και βουλευτές και από την αντιπολίτευση αλλά και από τη Γερουσία όπου υπάρχει, στην περίπτωση που υπάρχουν δύο ε, βουλές στα κράτη-μέλη. Επίσης ε, θα γίνεται συμπροέδρευση από την χώρα που θα έχει την εκπεριτροπής προεδρία του Συμβουλίου και από τον πρόεδρο της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Θέλουμε να επιμείνουμε στις ανεπάρκειες της πρότασης κανονισμού σε σχέση με την Ευρωπόλ που αναφέρθηκαν προηγουμένως ότι αφορά την προστασία των δεδομένων. Υπερθυμίστηκε αυτό, αλλά επιμένουμε εκ νέου καθώς δεν βλέπουμε να σημειώνεται πρόοδος ε, στο θέμα της προστασίας των δεδομένων. Επομένως πρέπει να επαγρυπνούμε σε σχέση με το τι μπορεί να προβλεφθεί μέσω αυτού του κανονισμού. Αυτή είναι προς το παρόν η θέση του Γαλλικού Κοινοβουλίου και σε ένα μήνα θα ολοκληρωθεί και θα γίνει η θέση της Εθνοσυνέλευσης ε, μετά την εξέταση από την Αρμόδια Επιτροπή. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ και πράγματι το εγγραφό σας έχει διανεμηθεί, νομίζω ότι το έχετε όλοι. Να διαβάσω τους επόμενους ομιλητές. Karsten from Denmark, then Mr. Alexander I hope, from Poland, then Mr. Brons, Θέλει κάποιο άλλο το λόγο, γιατί κατόπιν θα κλείσω τον κατάλογο των μιλτών. Ο κύριο Μισελ, ναι, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, και εγώ χαιρόμαι ιδιαίτερα που έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε εδώ με τους εκπρόσωπου των Εθνικών Κοινοβουλίων και φυσικά του καλωσορίζω. Με ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι συνεισφορές τους στη συζήτηση αυτή, γιατί είναι σημαντική συζήτηση και επί τη ουσία, αλλά ε, είναι και πραγματικά μας δείχνει και κάποιες παράξενες θέσεις. Ε, οι σκιώδες μας δεν είναι εδώ σήμερα, έτσι λοιπόν τον αντικαθιστώ. Φυσικά εμείς θέλουμε ενίσχυση της Ευρωπόλ για να είναι πιο αποτελεσματική, αλλά κυρία Ματιέ θέλουμε να είναι και πιο δημοκρατική η Ευρωπόλ, γιατί θα πρέπει να ασκείται δημοκρατικό έλεγχο σε αυτή την υπηρεσία. Όταν ακούω κάποια επιχειρήματα μου δημιουργούνται κάποιε ανησυχίε, δηλαδή να, να θεωρηθούν κάποιε συμφωνίε που έτυχαν δύσκολη ε, διαπραγμάτευση. Ε, δηλαδή, τι θα κάνουμε, θα κρυβόμαστε για να ζούμε ευτυχεί. Ε, Όμω αυτό δεν συνάδει με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ούτε με το κράτο δικαίου. Δεύτερον, δεν άκουσα και φυσικά ε, γνωρίζω τον πρίο του εισηγητή μας ε, και τον εμπιστεύομαι, όμως δεν άκουσα από την πλευρά του, τουλάχιστον μέχρι τώρα, κάποια επιχειρήματα που πράγματι να είναι ισχυρά για να μας δείξουν ότι μία συγχώνευση μεταξύ Επόλ και Ευρωπόλ θα μείωνε την προστιθέμενη αξία. Εγώ βλέπω όμως την προστιθέμενη αξία στη συγχώνευση γιατί όταν βλέπουμε ότι η Κομισιόν στην πρόταση της ε, προτείνει ε, να έχουμε μία ακαδημία στα πλαίσια της Ευρωπόλ όπου εκεί θα συνδυάζεται και η εμπειρία της Ευρωπόλ αλλά και η υλοποίηση των ε, κυρίων επιστολών με ένα τρόπο πολύ πιο σοβαρό. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν θα έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο και νομίζω ότι οι λόγοι για να μην γίνει είναι μάλλον συναισθηματική, ότι δεν χρειάζονται πάρα πολλέ μεταρρυθμίσει, να τα αφήσουμε όλα όπω έχουν, δεν είναι σημαντικέ οι συνέργειε, ούτε η οικονομία, ούτε ε, η συνοχή. Όμω ε, αυτά ζητάει η κοινή γνώμη στην Ευρώπη σήμερα και στη συνέχεια ξέρω το ποιόν ε, των ομιλητών. Έτσι λοιπόν δεν νομίζω ότι πίσω από αυτό κρύβεται κάποιος οπορτουνισμός ή ένα είδος ε, υπολογισμού. Εγώ νομίζω ότι αν υπάρχει ένα στοιχείο που μου φαίνεται συνεκτικό και ότι θα επέφερε προς τη αξία θα ήταν ε, η συγχώνευση αυτών των δύο υπηρεσιών δεν βλέπω καθόλου πού θα ήταν η προσθέμενη αξία στο να διατηρήσουμε τις δύο υπηρεσίε σε διάφορετικές τοποθεσίες. Η γιαγιά μου που ήταν αγρότησα δεν θα το είχε καταλάβει αυτό. Ούτε κι εγώ βέβαια το καταλαβαίνω. Αυτά ήθελα να σας πω. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Ξεπέρασα και το χρόνο, αλλά ξέρετε, είμαι παθιασμένος για το ζήτημα αυτό. Και δεν τοποθετήθηκα από της ουσίας, αλλά θα το πράξω στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Κάστανταβιτσον από τη Δανία. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να έρθω εδώ σήμερα και να σας εκφράσω τις απόψεις της Βουλής της Δανίας για το θέμα αυτό. Η Δανία έχει κάποιες ε, ιδιαιτερότητες όσον αφορά την Ευρωπόλη. Έχει το δικαίωμα opt-out σε ορισμένες ε, νομικές υποθέσεις. Θα πρέπει κάποτε να αλλάξει βέβαια αυτό, όμως μέχρι να γίνει αυτό και να διεξαχθεί το δημοψήφισμα βρισκόμαστε σε μια περίεργη θέση όσον αφορά την Ευρωπόλη και τους ε, μελλοντικού διακανονισμούς σχετικά με αυτή. Και το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν εξετάσει εντελεχώς, ε, βρίσκουμε την ε, πρόταση αυτή. Εμείς ε, δεν θέλουμε να απέχουμε για πάντα από αυτό, όμως θέλουμε να κρατήσουμε λίγη απόσταση. Τώρα, θα ήθελα να απαντήσω γραπτώς στα σχόλια που έχουν ήδη διατυπωθεί. Ορισμένοι έχουν ήδη αναφέρει το θέμα του κοινοβουλευτικού ελέγχου και τη μονάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου που θα συσταθεί. Αυτή η μονάδα χρειάζεται να είναι ευέλικτη και αποτελεσματική στον τρόπο εργασίας της. Επίσης πιστεύω πως αξίζει να σημειωθεί ότι τουλάχιστον κατά τη δική μας άποψη η ισορροπία που έχει επιφέρει αυτή η πρόταση και οι τροπολογίες ε, μας φαίνεται κάπως μας φαίνεται αρκετή, ικανοποιητική. Ε, ιδιαίτερα η πρόβλεψη για την κοινή Επιτροπή Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. Ε, βέβαια, στη Δανία έχουμε τρεις διαφορετικές επιτροπές που ασκούν τέτοιου είδους ελέγχους και δεν θα τέριαζε καλά στο δανεικό μοντέλο αυτή η πρόταση. Εμείς θα επιθυμούσαμε να δούμε καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην Επιτροπή ΛΥΜΠΑ και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Αυτό συμφωνεί και όλας και με την Ιρλανδική πρόταση που έχει διατυπωθεί γραπτός. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πόισετς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Στην Πολωνία η γνώμη είναι θετική για την ε, νομοθετική πρωτοβουλία που προβλέπει στον εξυγχρονισμό της νομικής βάσεως για την Ευρωπόλη και την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπόλη, Γνωρίζουμε την ανάγκη προσαρμογή τη νομική βάση στην συνθήκη της Λισαβόνα. Θεωρούμε ωστόσο ότι πρωτίστω πρέπει να γίνει προσπάθεια να βρεθούν λύσεις που να επιτρέψουν να προχωρήσουν, να εξυγχρονιστούν, να τελειοποιηθούν οι μηχανισμοί και όχι να ξαναρχίσουν όλα από την αρχή. Στην Πολωνία λέμε συχνά ότι το καλύτερο είναι εχθρός του καλού. Γι' αυτό τον λόγο μας ανησυχεί. Λίγο το σύνολο του προτάσεων που υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία στοχεύει σε μια σε βάθος αναδιάρθρωση των αστυνομικών συνεργασιών στην Ευρώπη. Θέλει να συγχωνεύσει την Ευρωπόλ με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία. Τώρα, για την ώρα, δεν βλέπουμε να υπάρχουν αποχρόντες λόγοι που να δικαιολογούν τέτοια συγχώνευση. Δεν βλέπουμε δηλαδή να διαμορφώνεται προστιθέμενη αξία ούτε σοβαρές εξοικονομήσεις που να ωφελήσουν τις χώρες μέλη. Δύο λόγια τώρα για την παρέμβαση της συναδέλφου από την Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Ίσως εννοεί τον κύριο Μισελ, γιατί μας μίλησε ο κύριο Μισελ για την γιαγιά του. Τώρα εμείς λέμε στην Πολωνία ότι κότες και γελάδες δεν πάνε μαζί. Εμείς πάντως είμαστε ικανοποιημένοι από τις άλλες προτάσεις για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Συμφωνώ με όσους μίλησαν προηγουμένως ότι ο έλεγχος πρέπει να διατηρηθεί στο υφιστάμενο πλαίσιο και να μην ανατεθεί σε νεοειδρυθισόμενα όργανα. Όπως άλλωστε είπαμε ήδη σήμερα, άλλος δηλαδή συνάδελφος, και εμείς σώμεθα υπέρ ενός ε, ελέγχου light που δεν θα αμφισβητήσει κάποιες δραστηριότητες της ε, Ευρωπόλ που απαιτούν κάποια διακριτικότητα και κάποιες εμπιστευτικές διαδικασίες. Μας ικανοποιούν επίσης οι προτάσεις για τους μηχανισμούς προστασίας ε, των προσωπικών δεδομένων που χειρίζεται η Ευρωπόλ. Εκεί τονίζουμε την ανάγκη να βρεθούν αποτελεσματικές λύσεις. Επαναλαμβάνουμε δηλαδή ότι θα πρέπει να είναι δυνατόν να συνδυαστεί η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης προσωπικών δεδομένων με την συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ενωτήτων και βεβαίως ιδίως με την εξασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπρόντς. Μάλιστα. Ακούσαμε ότι η Ευρωπόλ θα αποκτήσει μια νέα δυνατότητα ανταπόκρισης για το κυβέρνο έγκλημα και έχουν αναφερθεί ήδη ορισμένα ε, σημεία ή απάτη με τις επιστοτικές ε, κάρτες, αντιμετώπιση τρομοκρατίας και φυσικά κανείς δεν θα είχε αντίρρηση για ε, τις αποτελεσματικές μεθόδους που θα ήταν αναγκαίες έτσι και να καταπολεμηθούν αυτά τα εγκλήματα. Τώρα, εάν το κυβέρνο έγκλημα επεκταθεί και παρεμποδίζει ορισμένες ε, επικοινωνίες. Και εάν ε, η νομοθεσία ε, που είναι περιοριστική επεκταθεί και σε άλλες χώρες, αυτό θα ήταν κάτι που θα με ανησυχούσε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπρόντς. Εγώ απομένω ως τελευταία ομιλήτρια και θα Είμαι πειθαρχημένη όσον αφορά το χρόνο Τώρα έμαθα πως ε, κότες και γελάδες δεν πάνε στον ίδιο στάβλο. Βέβαια δεν ξέρω ποιες είναι οι κότες και ποιες είναι οι γελάδες. Θα είμαι σύντομη, όπως και να έχει, καταρχάς όσον αφορά την κοινή κοινοβουλευτική εποπτεία. Ναι, αλλά πρέπει αυτή να είναι αποτελεσματική. Και για να είμαι ειλικρινής, αν δημιουργήσουμε μια τέτοια επιτροπή από μέλη της Επιτροπής ΕΛΥΜΠΕ και μέλη ε, του κάθε κράτους εμέλους, θα καταλήξουμε με 116 βουλευτές. Και ειλικρινά δεν βλέπω πώς μπορούμε έτσι να διασφαλίσουμε μια αποτελεσματική εποπτεία με τόσους ε, πολλούς ανθρώπους. Εάν εγώ ήμουν διευθύντρια της Ευρωπόλ θα χαιρόμουν πάρα πολύ διότι θα είχα την ελευθερία να κάνω ό,τι θέλω. Δεν πρέπει ε, να μην έχουμε εμπιστοσύνη. Εντάξει, διακρίνω κάποια, κάποιον ανταγωνισμό εδώ και Επιτρέψτε μου να πω κάτι όχι για τους παρόντες αλλά για τους απόντες. Εδώ αντιπροσωπεύονται 7 κράτη-μέλη. Έχουν έρθει 7 κράτη-μέλη. Και ελπίζω πως οι υπόλοιποι θα έπρεπε να ήταν εδώ προτού καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα και θα έπρεπε να υπάρχει αρκετό περιθώριο λιγμών στην Ευρωπόλ. Εγώ θα προτιμούσα ε, ενδεχομένως στο τέλος η Ευρωπόλ να γίνει κάποιου είδους ε, αστυνομική αρχή. Όμως η ε, εποπτεία είναι προϋπόθεση, δεν είναι εμπόδιο για την επιχειρησιακή ελευθερία. Είναι προϋπόθεση. Και μάλιστα οι πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με την κατασκοπία από τις κυβερνήσεις έχουν δείξει την ανάγκη για περισσότερη δημοκρατική εποπτεία και όχι λιγότερη. Τώρα, όσον αφορά τις τροπολογίες που έχω συνυπογράψει για την ε, εποπτεία και την επίβλεψη όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Πιστεύω και απευθύνομαι προς τον εισηγητή ότι χρειάζεται μια αποτελεσματική εποπτεία, αποτελεσματικός έλεγχος και γι' αυτό και υποβάλαμε αυτές τις τροπολογίε. Υπήρξε βέβαια κάποιο ε, φόβο. και τέλος να πω ότι υποβάλαμε μια τροπολογία που ίσως είναι κάπως αμφιλεγόμενη, που ζητά αρμοδιότητε τη Ευρωπόλη έτσι ώστε αυτή να διερευνά τι ε, μεγάλη κλίμακα κλίμακας ε, και να αναλαμβάνει αν χρειάζεται πρωτοβουλία. Και αυτό το υποβάλαμε έχοντας υπόψη αυτό που έγινε στους σερβερς της SWIFT στην Ολλανδία και εκεί η κυβέρνηση αρνήθηκε να ερευνήσει και αυτό είναι κάτι που επηρέασε το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπόλη, λοιπόν θα έπρεπε να έχει τις αρμοδιότητες να διεξάγει έρευνες εκ μέρους της Ένωσης. Επίσης ε, με αυτό να πω ότι τελείωσα. Έχουμε 27 λεπτά ακόμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διεξάγουμε ένα δεύτερο κύκλο συζητήσεων. Εάν κάποιος από εσά έχει έτσι νιώθει την ανάγκη να κάνει κάποια σχόλια σχετικά με τα όσα υπόθηκαν, τότε παρακαλώ να το κάνει. Ο Λόρδε Χάνεϊ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που μου ξαναδίνετε το λόγο. Ελπίζω να μην κάνω κατάχρηση του σε αυτή τη φορά. Είναι κρίμα, πιστεύω, που δεν έχουμε καταφέρει να κοιτάξουμε περισσότερο τι γίνεται με την εντολή για την μονάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου που έχει προταθεί, διότι αυτή η μονάδα είναι κάτι που εγώ και η Επιτροπή μου θεωρούν αρκετά προβληματικό σημείο. Όσον αφορά το σχολείο σας για το μέγεθος της Επιτροπής αυτής, υποθέτω πως έχετε δίκιο. Εάν τα εθνικά κοινοβούλια αποκτήσουν ικανοποιητικά ικανοποιητικέ θέσει εμελών, ε, τότε όντω ο αριθμό ε, των εμελών θα είναι πολύ μεγάλο. Όμω ε, δεν πρέπει να είναι πολύ μικρό έτσι κι αλλιώ. Πιστεύω λοιπόν πως είναι καλύτερο να ε, συνεχίσουμε έτσι. Θα είναι περισσότερο κοινοβουλευτικός ο χαρακτήρας και όχι κατά περίπτωση, αλλά όπως έχουν πει ήδη και άλλοι ομιλητές, δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικά παρεμβατικοί στην άσκηση ελέγχων, ε, δημοσιονομικών ελέγχων. Υπάρχουν εξάλλου και άλλοι μηχανισμοί που προβλέπουν ελέγχους. Γι' αυτό λοιπόν και θα ήθελα να τονίσω αυτό το σημείο. Κυρία Έρνστ, έχετε το λόγο. Ε, είναι καλό το ότι συνεχίζουμε τη συζήτηση. Γιατί για να είμαι σε βλέπω ότι κάθε εθνικό κοινοβούλιο αναφέρεται στο τι γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο, στο πώς διεξάγονται οι έλεγχοι από την αστυνομία. Και αυτό που διαφαίνεται είναι ότι οι αρμόδιοι παντού επιθυμούν να ελαχιστοποιηθεί ο έλεγχος και αυτό πιστεύω πως δεν πρέπει να αφήσουμε να επιτραπεί. Χρειάζεται ένας αποτελεσματικός έλεγχος και πιστεύω πως αυτή εδώ η Επιτροπή, η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, ήδη έχει αρκετές αρμοδιότητες και ικανοποιητικά αποτελέσματα. Υπάρχουν πάρα πολλές ε, επιτροπές ε, οι οποίες ε, συνεργάζονται και εγώ θα προτιμούσα πολύ περισσότερο και θα φερούσα εξάλλου και πολύ ε, σωστότερο να υπάρχει ε, η δομή έτσι όπως είναι. Φυσικά και χρειαζόμαστε διαβούλευση και ανταλλαγή απόψε με τα εθνικά κοινοβούλια, οπωσδήποτε. Ε, χρειάζεται να συζητήσουμε για ε, όσα έχουν να κάνουν με το συντονισμό, βέβαια. Αλλά πιστεύω πως αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα, διότι δεν μπορώ να καταλάβω πώς με τόσους σε πολλούς ανθρώπους θα καταφέρουμε να έχουμε έναν αποτελεσματικό έλεγχο και πώς το κάθε κράτος μέλος θα το επιτύχει αυτό. Μόνο και μόνο την νομική βάση πάρτε. Εγώ πραγματικά δεν θέλω να υπάρχει κάποιο εδώ που θα είναι εδώ και θα κάθεται και θα μου λέει πω ε, δεν είναι ευχαριστημένο μαζί μου. Αυτό δεν είναι έλεγχο, αυτά είναι αστεία πιστεύω. Γι' αυτό και θεωρώ πώ πρέπει να δούμε ακριβώ το πρόβλημα. Ναι, θέλουμε να υπάρχει έλεγχο, αλλά πρέπει να δούμε πώς θα γίνεται αυτός ο έλεγχος σε μεμονωμένες ε, περιπτώσεις. Ε, εγώ δεν πιστεύω πώ Θα γινεται αυτό ο έλεγχο σε μεμονωμένε περιπτώσει. εγω δεν πιστευω μαζί μας όλοι και δεν πρέπει να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να καταλήξουμε έτσι. Ευχαριστώ πολύ και στο τον κύριο Χόλτσε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Παρανόηση, να αποφύγουμε παρανόηση ότι ενδεχόμενα έλεγχος σημαίνει και παρέμβαση στο επιχειρησιακό μέρος των λειτουργιών της Ευρωπόλ. Εγώ απλώς εννοώ ότι ανα πάσα στιγμή μπορούμε να ζητήσουμε πληροφορίες. Δεν σημαίνει ότι πάμε να φτιάξουμε ένα έξτρα διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπόλ. Επανέρχομαι στην ε, παρέμβαση του Λόρδου Χάνε. Είναι σημαντικό να συμμετάσχουν όλα τα κοινοβουλευτικά σώματα. Στι διάφορε χώρε μέλη υπάρχουν διαφορετικές κοινοβουλευτικές παραδόσεις, ορισμένες με δύο κοινοβουλευτικά σώματα. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Γενικά πάντως θεωρώ ότι η συζήτηση αυτή πρέπει να διεξαχθεί ακόμα περισσότερο σε βάθο. Για μένα πάντως ο έλεγχος αποτελεί σημαντική προϋπόθεση. Και εφόσον με τον τρόπο αυτό ε, δημιουργηθεί εμπιστοσύνη, τότε θα μπορέσει να δράσει και όλας ο οργανισμός αυτός πιο αποτελεσματικά. Άλλος κανείς θέλει να λάβει ξανά το λόγο πριν επανέλθουμε στον εισηγητή, αλλά θα πω εγώ δύο λόγια, διότι σωστά είπατε ότι υπάρχει ανάγκη για πρόσβαση σε έγγραφα και μεγαλύτερη διαφάνεια κλπ. Και ο αναθεωρημένος κανονισμός, για, η αναθεώρηση μάλλον του κανονισμού για την πρόσβαση στα έγγραφα έχει κολλήσει στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν. Αυτά τα πράγματα ωστόσο συμβαδίζουν. Διαφάνεια και πρόσβαση σε έγγραφα είναι σημαντικά στοιχεία κλειδιά για οποιαδήποτε έννοια δημοκρατικής υποπτίας. και βεβαίως γνωρίζουμε τα προβλήματα που έχουν προκληθεί από την άρνηση της Ευρωπόλου να επιτρέψει πρόσβαση σε έγγραφα. Ε, γνωρίζω και εγώ επειδή συμμετέχω σε ε, προσφυγές και ενώπιον του Ευρωπαίου Συνηγόρου του Πολίτη για σχετικά θέματα. Έχουμε το ενδιαφέρον λοιπόν, αλλά και εσείς ως εθνικοί βουλευτές για τον αναθεωρημένο. Να εγκριθεί δηλαδή το συντομότερο δυνατόν ο αναθεωρημένος κανονισμός για την πρόσβαση έγγραφα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ας επιστρέψω τώρα. Α, με συγχωρείτε μια στιγμή. Έχω ακόμη μια τελευταία παρέμβαση της κυρίας Καραμαλή. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επανέλθω στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και στην εκπροσώπηση των Εθνικών Κοινοβουλίων. Άκουσα την επιθυμία σας να μην ε, είναι πολυπληθής αυτή η Επιτροπή, αυτό, αυτή η μονάδα ελέγχου. Όμως, ε, καθώς ε, προτείνονται δύο μέλη για κάθε κοινοβούλιο, αν αυτό σας φαίνεται υπερβολικό, τότε τουλάχιστον θα έπρεπε να έχουμε ένα βουλευτή ε, ανακοινοβούλιο γιατί δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τη γερουσία ε, από τις, στις χώρες στις οποίες υπάρχει. Θα πρέπει λοιπόν ε, όλες οι εθνοσυνελεύσεις να μπορούν να συμμετέχουν ε, σε αυτή τη μονάδα ακόμη και αν λάβουμε υπόψη ότι μπορεί να υπάρχει και κάποιο αναπληρωτή που θα μπορεί να αντικαταστήσει του διορισμένου συναδέλφου. Μάλιστα, ευχαριστώ. Τώρα ερχόμαστε στον εισηγητή, ο οποίο ε, θα πρέπει να καταφέρει να μας παρουσιάσει τις κατάλληλες λύσεις έτσι ώστε να εκπροσωπηθούν σωστά τα εθνικά κοινοβούλια και όσα έχουν ε, ένα σύστημα με δύο εθνοσυνελεύσεις. Εγώ νομίζω ότι ο κ. Δεμέρα είναι πολύ ικανός για να επιτελέσει αυτό το καθήκον. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για τα ευγενικά σου λόγια. Εγώ θέλω να κάνω μία σύνοψη των 20 ε, παρεμβάσεων που ακούσαμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Ε, η σύνοψη μπορεί να καλύψει τρεις πτυχές. Το θέμα της συγχώνευσης, το θέμα της μονάδας κοινοβουλευτικού ελέγχου και το θέμα της ανησυχίας που εκφράστηκαν για τις εγγύσεις προστασίας των δεδομένων σε μια υπηρεσία ασφαλείας. Εγώ θα ήθελα να προβούσω μια προσωπική εξομολόγηση εδώ. Εγώ ήμουν ε, και ελεγκτής, αλλά και ήμουν και αντικείμενο ελέγχου. Έχω συμμετάσχει και στο Εθνικό Κοινοβούλιο και στην Γερουσία και είχα και αρμοδιότητε στη χώρα μου για θέματα ασφαλείας. Επίσης, σε άλλο στάδιο της ζωή μου ήμουν και μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπόλου. Επομένω, ε, δεν ε, γνωρίζω τα θέματα αυτά μόνο στη θεωρία. Και όταν ε, έκανα την νομοθετική μου πρόταση, στάθμισα πάρα πολύ τις αρμοδιότητες ελέγχου που έχουν τα Εθνικά Κοινοβούλια επί των ε, αστυνομικών τους αρχών και των υπηρεσιών τους ασφαλείας. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι αρμοδιότητες των Εθνικών Κοινοβουλίων ε, σε σχέση με τον έλεγχο της αστυνομίας είναι πολύ μεγαλύτερες από τις αρμοδιότητες που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον έλεγχο της Ευρωπόλ. Και πρέπει να πούμε στη συνέχεια πως οι αρμοδιότητες της Ευρωπόλ είναι πολύ μικρότερες από τις αρμοδιότητες που έχουν ε, οι αστυνομικές αρχές στα κράτη-μέλη. Λοιπόν, αυτό είναι το περιτύλιγμα. Θα μπω τώρα στο περιεχόμενο. Γνωρίζετε και αν όχι θα έπρεπε να γνωριστε ότι εδώ και τρία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μπορεί να μας το διαβεβαιώσει η κυρία Νταμίτση εργάζεται για την προετοιμασία αυτής της νομοθετικής πρότασης και σε αυτό την ίδια αίθουσα συζητήσαμε μια ολόκληρη ημέρα με τους εκπροσώπους των Ενδρικών Κοινοβουλίων το θέμα του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Επομένως, οι ιδέες μου που αντικατοπτρίζονται στη μονάδα ελέγχου, που θα μπορούσε να ονομαστεί και με άλλο τρόπο, οι ιδέες μου αποτελούν συνέπεια και συνθετικού έργου των συζητήσεων αυτών που έχουν λάβει χώρα τα τελευταία τρία χρόνια και έχουν συμμετάσχει στις συζητήσεις αυτές αναμφισβήτητα και τα Εθνικά Κοινοβουλία και φυσικά και η Βουλή των Λόρδων. Όταν εγώ λοιπόν προτείνω τη δημιουργία αυτής της μονάδας ελέγχου, μιλώ για την ανάπτυξη του άρθρου 88 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο αυτό για να καθησυχάσω τον ε, κύριο Κίρκοφ, ε, τον οποίο θαυμάζω, αυτό το άρθρο 88 δίνει ασφάλεια δικαίου στη μονάδα ελέγχου και ασφάλεια δικαίου προσδίδει και η συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων και το λέει κατηγορηματικά το άρθρο 88. Δεν υπάρχουν αμφιβολίες λοιπόν. Τώρα, η μονάδα ελέγχου που είναι απαραίτητη, έχει δίκιο ε, η Σοφή, θα πρέπει να είναι μικρή αυτή η μονάδα και εξειδικευμένη για να είναι αποτελεσματική. Και να πω στην συνάδελφο από την Γαλλία, στη δική μου πρόταση, λέω ότι πρέπει να υπάρχει ένας εκπρόσωπος από κάθε εθνικό κοινοβούλιο, ένας εκπρόσωπος που θα είναι εξειδικευμένος από την αμόδια επιτροπή του Εθνικού Κοινοβουλίου θα προέρχεται. Γιατί αν έχουμε δύο νομίζω ότι θα είναι υπερβολικός ο αριθμός. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα καθήκοντα της μονάδας ούτε καν ε, διανοούμαστε να εμπλέκει σε έρευνες ή να ζητά πληροφορίες που αφορούν μια έρευνα. Σε καμία περίπτωση εδώ, όταν ε, μιλάμε για το SWIFT ή για τα PNR, τα δεδομένα καταλόγου των επιβατών, πρέπει να εξετάσουμε κάποια έγγραφα που είναι απόρριτα, είναι διαβαθμισμένα και υπάρχουν πολύ μεγάλες εγγύσεις, μπαίνει το έγγραφο στην αίθουσα, μόνο οι βουλευτές μπορούν να το δουν και κατόπιν επιστρέφεται, δεν βγάζουμε φωτοτυπίες, τίποτα. Επομένως, ξέρω πολύ καλά για τι πράγμα μιλάω και σταθμίζω όλες τις δυνατότητες στον τομέα του ελέγχου, όμως είναι απαραίτητος εντελώς απαραίτητος ο κοινοβουλευτικός έλεγχος και μάλιστα ενισχύει την Ευρωπόλ και τις προσδίδει ασφάλεια δικαίου. Και ένα μικρό σχόλιο για τον κύριο Μίτσελ, τον οποίο επίση θυμάζω. Εγώ για τον κύριο Μισελ. Εγώ είμαι εντελώς αντίθετος για τη συγχώνευση και ξέρω ότι η φιλελεύθερη είναι υπέρ. Όμως τώρα εδώ δεν θέλω να κουράσω τους συναδέλφους. Ε, εγώ σας διαβεβαιώ ότι αυτά τα επιχειρήματα που είναι κατά της συγχώνευσης είναι πάρα πολύ λογικά. Άλλο σχόλιο για τον συνάδελφο από την Ουγγαρία. Όπως και η Ουγγαρία και εμείς είμαστε κατά της συγχώνευσης. Όμως, είμαστε και κατά του τρόπου που χρησιμοποίησε το Συμβούλιο, ε, του διαστραμμένου τρόπου που χρησιμοποίησε το Συμβούλιο για την εφαρμογή των συνθήκων. Ακατάλληλα, ιδιαίτερα ακατάλληλα, χρησιμοποίησε το Συμβούλιο το άρθρο 341, που είναι αυτό το οποίο αναφέρεται στις έδρες και στην ικανότητα του Συμβουλίου να διορίσει τις έδρες, να καθορίσει τις έδρες. Το 341 μιλά για τους θεσμούς, για τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο θα μιλήσουμε για ένα θεσμό και την έδρα του, στην Ολομέλεια, για την έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όμως μια υπηρεσία δεν είναι θεσμός, θεσμός είναι το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο, Κομισιόν. Το 341 δεν εφαρμόζεται λοιπόν εδώ. Και καθώς έχουμε αυτές τις αμφιβολίες, γι' αυτό ζητήσαμε μία γνωμοδότηση από την νομική υπηρεσία, η οποία θα πρέπει να παρουσιαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφού παρουσιαστεί θα αποφασίσουμε ποια οδό θα ακολουθήσουμε και τι θα κάνουμε. Όμως, προς στιγμή ναι, δεν έχουμε να πούμε τίποτα σε σχέση με τι έδρε, Γιατί η νομική βάση δεν είναι η αρμόζουσα και αφού έχουμε και την γνωμοδότηση νομική υπηρεσία, θα τοποθετηθεί η Επιτροπή μα σχετικά με το θέμα αυτό. Τρίτο σημείο και τελευταίο κυρία Πρόεδρε, η προστασία των δεδομένων. Για μας είναι πολύ σημαντική η προστασία των δεδομένων εντός μιας υπηρεσίας ασφαλείας. Γιατί? Γιατί εγώ ίδιος το ομολογώ και σας ζητώ συγγνώμη αν το πάρετε ως ματαιόδοξο το σχόλιο. Εγώ ιδιώς ε, εδώ και τρία-τέσσερα χρόνια από τότε που ήμουν εισηγητής για την απόφαση συμβουλίου έχω ζητήσει τη συμμετοχή του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασία του Δεδομένου του κ. Χάστινγκ και όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία των δεδομένων εντό τη Ευρωπόλ. Και αυτό ακόμη και αν έχει να κάνει με την κοινή αρχή ελέγχου. Μιλώ για τις εγγυήσεις που πρέπει να εφαρμόζονται σε μια υπηρεσία ασφαλείας. Και στις 26 του μήνα θα συναντηθώ εκ νέου με τον κύριο Χάστινγκ για να τον ενημερώσω σχετικά με την πρόοδο των εργασιών μας και επειδή και ο κύριος Χάστινγκ θέλει να συναντηθεί και να συνομιλήσει μαζί μου, επειδή ε, τώρα εδώ είμαστε εντελώ βυθισμένοι στην οδηγία και στον κανονισμό προστασίας των δεδομένων και θέλουμε να εφαρμόσουμε αυτή την νομοθεσία σε μια υπηρεσία ασφαλείας. Επομένως, ε, εμείς λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις ενισφορές των Εθνικών Κοινοβουλίων, θα λάβουμε υπόψη όλα τα έγγραφα που θα μας σταλούν, αλλά εμείς έχουμε την ικανότητα να νομοθετούμε, αλλά εσείς έχετε την δυνατότητα να επηρεάσετε τους νομοθέτες και εμείς ευχαριστώ σταφεθούμε σε αυτή την επιρροή γιατί τη χρειαζόμαστε, τη θέλουμε αυτή την επιρροή. Γιατί όχι μόνο για την επιτακτική νομοθετική ανάγκη που προέρχεται από την συνθήκη της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και επειδή θέλουμε η Ευρωπόλ να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική και να έχει και έναν κοινό έλεγχο από τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σιγητή. Στο τέλος αναφερθήκατε στην προστασία προσωπικών δεδομένων και τον ε, κανονισμό η οδηγία να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε μια έκκληση στους συναδέλφους μας από τα Εθνικά Κοινοβούλια να πιέσουν τις κυβερνήσεις τους να υιοθετήσουν την οδηγία ιδιαίτερα ε, όσον αφορά την ε, επιβολή του νόμου και να το κάνουν σύντομα χωρίς καθυστερήσεις για να μην καθυστερήσει και η διαδικασία. Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος αυτού του σημείου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια θερμότατα για την παρουσία τους. Ε, απόλαυσα πολύ την ανταλλαγή απόψεων και πιστεύω πως ε, αυτή διεξήχθη με πνεύμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Ελπίζω να έχουμε και άλλες συζητήσεις στο μέλλον, τέτοιου είδους και να βρούμε καλές λύσεις υπό την καθοδήγηση του εισηγητή μας φυσικά. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε λοιπόν. Διακόπτεται η συνεδρίαση για 8 λεπτά μέχρι τις 11.30. Αλλά μόλις μου λένε πως όλοι είστε παρόντες. Όσοι τέλος πάντων πρέπει να είστε εδώ. Σε αυτή την περίπτωση περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης η έκθεση του συναδέλφου Κάρλος Κοέλιο για την παρακολούθηση των εξωτερικών συνόρων στα πλαίσια της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα εσωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ένωσης. Κάποιος πρέπει να κάνει κάτι με τους τίτλους. Διαβάζεις έναν τίτλο και συνειδητοποιεί πόσο γελίο ακούγεται. Μία ολόκληρη πρόταση όπου τρεις φορές επαναλαμβάνεται επιχειρησιακή συνεργασία. Αστείο είναι αυτό. Συνάδελφοι, θα ήθελα να συζητήσω να καταλήψετε την αίθουσα ήσυχα και να συζητήσετε έξω από αυτή. Σας ευχαριστώ. 170 Λοιπόν, τροπολογίες υποβλήθηκαν ε, για την έκθεση του κυρίου Κοέλιο και πρώτα θα δώσω το λόγο στον ίδιο έτσι ώστε να τις σχολιάσει και μετά θα ζητήσω από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να παρέμβουν και έπειτα θα αρχίσει η συζήτηση, θα ανοίξει η συζήτηση για τα υπόλοιπα μέλη. Κύριε Κοέλιο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου, ιδιαίτερα τους κοιόδης εισηγητέ για τη συνεισφορά του. Πρέπει να πω ότι όταν κοίταξα τις ε, τροπολογίες ε, δεν είχαν έρθει όλες οι μεταφράσεις, αλλά από αυτά που βλέπω οι τροπολογίες χωρίζονται σε τρία Ήδη τρεις κατηγορίες, εκείνες που θέλουν να περιορίσουν το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού και να περιορίσουν τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό. Και όπως καταλαβαίνετε δεν μπορώ να τις δεχτώ εκείνες οι τροπολογίες που θέλουν να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού και τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά το γεγονός ότι θα θέλαμε να το κάνουμε δεν μπορούμε και τέλος αρκετές τροπολογίες οι οποίες πραγματικά συνεισέφεραν πολύ θετικά στην έκθεση και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που τις υπέβαλε λάβαμε περίπου 200 τροπολογίες. Γι' αυτό και πιστεύω πως ε, θα ήταν δίκαιο να ξανασυναντηθώ με τους σκιώδες εισηγητές έτσι ώστε να βρούμε κάποιους συμβιβασμούς για να γίνει πιο εύκολη η ψηφοφορία και να προσπαθήσουμε με τις συμβαστικές αυτές τροπολογίες να διατηρήσουμε την ισορροπία που προσπάθησα να έχω στην έκθεση. Εάν μου επιτρέπετε τώρα θα ήθελα να τονίσω πέντε σημεία τα οποία θεωρώ πως είναι τα κυριότερα στοιχεία της έκθεσης αυτής και των τροπολογιών, έτσι και αλλιώς. Καταρχάς, η νομική βάση. Εδώ μιλάμε για θαλάσσια παρακολούθηση και στα πλαίσια αυτά ε, μιλάμε για την ανάγκη να έχουμε σαφείς κανόνες όσον αφορά την ε, διάσωση, την αναζήτηση μόνο σε επιχειρήσεις που ε, συντονίζει η Frontex δηλαδή σε επιχειρήσει που συντονίζονται και χρηματοδοτούνται από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Οτιδήποτε πέρα από αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό νομικά. Πρέπει να δεχτούμε ότι ακόμα και αν ορισμένοι από εμάς θα ήθελαν να πάνε ένα βήμα παραπέρα, δεν είναι δυνατόν. Οφείλουμε να σεβόμαστε τι αρμοδιότητε των κρατών μελών, όπω και τα κράτη-μέλη οφείλουν να σέβονται τι αρμοδιότητε που έχουν δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας υπενθυμίσω επίσης ε, την δημιουργία ενός ε, χώρου δικαιοσύνης, η οποία δημιουργία χρειάζεται μια κοινή προσέγγιση και κοινή διαχείριση. Και αυτό δεν συμπεριλαμβάνει μόνο την ύπαρξη ενός επαρκούς ε, ελέγχου των εξωτερικών συνόρων, αλλά και τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες. Ωστόσο, η ανάγκη προστασία των συνόρων μας και η ανάγκη ύπαρξης ενός αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου των συνόρων πρέπει να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών που φτάνουν στα εξωτερικά σύνορα. Το δικαίωμα στη ζωή, τον σεβασμό, τα θεμελιώδη δικαιώματα και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίσουν πλήρη εφαρμογή αυτών. Επίσης, επόμενο σημείο που θα ήθελα να τονίσω, κυρία Πρόεδρε, είναι η ανάγκη σαφών κανόνων που θα ε, αφορούν την, τον κίνδυνο αποβίβασης. Γιατί χρειαζόμαστε αυτούς τους κανόνες. Αρκετά κράτη-μέλη επιχειρηματολογούν λέγοντας ότι δεν χρειαζόμαστε σαφείς κανόνες. Εγώ θα ήθελα να σας θυμίσω την κριτική που έχει ασκηθεί στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ε, της Frontex και τα ερωτήματα που έχουν δημιουργηθεί όσον αφορά την διάσωση από τη θάλασσα. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2010 ε, ψήφισε την απόφαση 252 για παρακολούθηση των θαλάσσιων συνόρων συντονισμένη από τη Frontex. Όπως ξέρετε αυτή η, αυτή η απόφαση έχει καταργηθεί με βάση την χάρτα των ε, δικαιωμάτων ε, δικαιοσύνης και εμείς έχουμε τώρα ως έργο να δημιουργήσουμε τους κατάλληλους κανόνες έτσι ώστε να διευκολύνεται το έργο της Frontex και το έργο αυτό να ε, συμμορφώνεται πάντα με τα πρότυπα για τα θεμελιώδη δικαιώματα και η, ε, να υπάρχει λογοδοσία από την αρμόδια Επιτροπή Συντονισμού. Το τέταρτο σχόλιο μου έχει να κάνει με περισσότερη αλληλεγγύη και με το να σωθούν ζωές. Τα ε, νότια θαλάσσια σύνορα της Ευρώπης, τη Μάλτα, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία, είναι τα σύνορα τα οποία έχουν να αντιμετωπίσουν τις πιο συχνές ε, αφήξεις διαθαλάσσης. Και παρά το γεγονός ότι αυτό το φαινόμενο δεν ε, έχει εξαπλωθεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, την επηρεάζει. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε περισσότερες κλήσεις για αλληλεγγύη και ανταπόκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να στηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτές τις χώρες οι οποίες επλήττονται περισσότερο από τις αφήξεις ε, δια της θαλάσσιας οδού. Η ανάγκη λοιπόν για αλληλεγγύη έχει γίνει απαραίτητη έτσι ώστε να διασφαλιστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των ε, μεταναστών αυτών τα πρόσφατα τραγικά συμβάντα στη Λαμπεντούσα, όπου χάθηκαν ανθρώπινες ζωές παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της ακτοφυλακής και των ενόπλων δυνάμεων της Μάλτας, να βοηθήσουν τα σκάφη αυτά που εξέπεμψαν σήματα κινδύνου, ε, έδειξαν ότι χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση των υφιστάμενων μηχανισμών έτσι ώστε να ε, είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην πρόληψη τέτοιων ε, ατυχημάτων στη θάλασσα. Ωστόσο, η κυβέρνηση της Ιταλίας, η οποία ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ψηφίσει ένα σχέδιο δράσης για το θέμα αυτό και ο Πρωθυπουργό της Μάλτας, ο οποίος ζήτησε, ο οποίος αναφέρθηκε σε νεκροταφείο στη Μεσόγειο, ζήτησαν δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη όμως τα δύο αυτά κρατημέλη μαζί με τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ελλάδα και την Κύπρο μπλοκάρουν την πρόταση αυτή η οποία περιλαμβάνει σαφείς κανόνες για την αναζήτηση και διάσωση μεταναστών, για τον ε, μόνο λόγο ότι αρνούνται να εφαρμόσουν οποιουσδήποτε ευρωπαϊκούς ε, κανόνες που αφορούν ε, την προστασία της ζωής των μεταναστών. Επίσης, άλλο σχόλιο έχει να κάνει με τους διεθνείς κανόνες αναζήτησης και διάσωσης μεταναστών και σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Όπως ξέρετε, το σχέδιο κανονισμού που εξετάζουμε τώρα ενώνει μέσα σε ένα νέο νομικό ε, μέσο τις υφιστάμενες διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του διεθνούς δικαίου που στοχεύουν να ξεπεράσουν τις διαφορετικές ε, ερμηνείες ε, της αναμοθεσίας που έχουν τα κράτη-μέλη και να αποφύγουμε τις αποκλίνουσες πρακτικές, να εξασφαλιστεί η σαφήνεια και ο σωστός συντονισμός των δράσεων από την Frontex. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου C355N μεταξύ άλλων λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρμόδια να δράσει στα πεδία που καλύπτει η απόφαση 2010 502. Επίσης είναι σαφές ότι το πεδίο εφαρμογής της πρότασης δεν υπερβαίνει την ε, ε, απόφαση του Συμβουλίου. Τα έξι κράτη-μέλη που ανέφερα μπλοκάρουν λοιπόν την πρόταση, η οποία περιέχει ξεκάθαρους κανόνες όσον αφορά την αναζήτηση, διάσωση και αποβίβαση των μεταναστών, ακόμα και αν περιορίζεται μόνο σε περιπτώσεις όπου ε, οι αρμοδιότητες αυτές ε, είναι μόνο συντονιστικές. Το άρθρο 10 για την αποβίβαση είναι, το, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς κανόνες της πρότασης ε, όσον αφορά τον, ε, την ε, διάσωση ανθρώπινων ζώων και την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τα κύρια επιχειρήματα που προέταξαν τα κράτη-μέλη αυτά για να στηρίξουν τη θέση τους ήταν τα ακόλουθα και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στα δύο κυριότερα επιχειρήματα. Το πρώτο λοιπόν είναι η έλλειψη αρμοδιοτήτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα που έχουν να κάνουν με αναζήτηση και διάσωση σε περίπτωση αποβίβασης. Να είμαι σαφής εδώ. Οι συνθήκες δίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την δυνατότητα να αναπτύξει μια συντονισμένη και κοινή μεταναστευτική πολιτική. Και εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια τέτοια αρμοδιότητα να ψηφίζει κανόνες για ελέγχους που θα αφορούν την ε, την, ε, τους, ε, ε, τους μετανάστες δεν θα εφαρμόζονται όταν αυτοί είναι υπό την εποπτεία των, της ακτοφυλακής. Δεν υπάρχει τίποτα στις συνθήκες που δίνει την δυνατότητα ελέγχου των ερευνών. Ωστόσο, ο στόχος του σχεδίου κανονισμού δεν είναι αυτός. Ο στόχος ε, σκοπεύει μόνο να ε, ρυθμίσει ε, την αναζήτηση και διάσωση μόνο στα πλαίσια της υφιστάμενης πολιτικής και τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μόνο σε περίπτωση που οι έρευνες αυτές συντονίζονται από την Frontex και που οι έρευνε αυτέ αφορούν μόνο την αναζήτηση και διάσωση σκαφών που έχουν εκπέμψει σήμα κινδύνου. Επίση, πιστεύουμε πω θα ήταν παράλογο να πιστεύει κανεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έχει ε, την ε, εξουσία να δημιουργεί προποθέσει Εφόσον η Frontex είναι μια υπηρεσία που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον ευρωπαϊκό ε, προϋπολογισμό. Το δεύτερο κύριο επιχείρημα από τα κράτη-μέλη, από αυτά μάλλον τα έξι κράτη-μέλη, είναι η συμβατότητα με το διεθνές δίκαιο το σχέδιο κανονισμού αναφέρεται ρητά στην συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο. Ε, χρησιμοποιείται η ίδια ορολογία, η οποία έχει γίνει ήδη δεκτή από τα κράτη-μέλη ε, σε νομοθεσία για την ενόμιμη μετανάστευση και τους συνοριακούς ελέγχους. Τώρα υπάρχει μια συμβατότητα και πιστεύουμε πως ε, είναι μόνο θέμα πολιτικής εθέλησης. Τώρα, όσον αφορά τις πιθανότητες αλληλεπικαλύψεων, δεν θα είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση ψηφίζει νομοθεσία η οποία ε, παρουσιάζει επικαλύψεις με την εθνική νομοθεσία, σκοπεύοντας ε, στην αποτελεσματική εφαρμογή ε, του, του, του νομικού πλαισίου. Τώρα, θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέκαθεν ήταν περήφανη για την πρωτοπόρο θέση της ε, ως υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ως ε, τέτοια. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτό αλλά και να συνεχίζουμε ε, με την προστασία των θεμελιωδών αυτών δικαιωμάτων. Τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να συνεχίσουν να έχουν μια τέτοια θέση και ε, πραγματικά θα ήταν αδύνατο να περασπιστούν μια τέτοια θέση η οποία ε, θα αρνείται την ευθύνη της να αναλάβει σαφή μέτρα έτσι ώστε να αποφευθούν οι πολύ άριθμοι θάνατοι στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης στα λεγόμενα νεκροταφεία της Ευρώπης στη Μεσόγειο Θάλασσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι... Μιλήσατε για κάποια υπερηφάνεια κύριε Σιγητά. Εμείς είμαστε υπερηφανοί για σας. Θα δώσω το λόγο τώρα στους και οδησηγητές, αν και δεν έχουν ακόμη ζητήσει όλοι το λόγο. Α, σωστά μου θυμίζεις ότι πρώτα πρέπει να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Προεδρία του Συμβουλίου, αλλά παρακαλώ να είναι πραγματικά πολύ σύντομη μέσα και στο πνεύμα της προηγούμενης συνάντησης, ε, συνεδρίασης. Ο κ. Νίλσεν, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να πω λίγα λόγια για τη συζήτηση αυτή σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες για το πεδίο εφαρμογής. Εκεί δεν έχω να προσθέσω πολλά στα όσα ήδη ανέπτυξε ο κ. Σκοέλιο και για την δυνατότητα ή μάλλον την έλλειψη δυνατότητας να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού καθώς και την καθαρή αρμοδιότητα που υπάρχει για τον ίδιο τον κανονισμό. Δεν έχω να προσθέσω εκεί τίποτε άλλο. Ορισμένες τροπολογίες τώρα έχουν ε, υποβληθεί για τα safeguard, για την αρχή των θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων στο άρθρο 4. Εκεί ε, είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την διάταξη. Βέβαια, οι κανόνες που θα θεσπιστούν θα πρέπει και να είναι δυνατόν να εφαρμοστούν στην πράξη και να είναι και οριζόντια εφαρμόσιμοι σε όλα τα σύνορα στις διάφορες όμορες χώρες και βέβαια και στο προσεχές μέλλον. Για τις τροπολογίες που έχουν σχέση τώρα με δυνατότητες ε, αναχέτησης, προσώπων που δεν βρίσκονται σε κατάσταση επίγουσα, δηλαδή που βυθίζονται τα σκάφη, αλλά που μπορεί να έχουν σχέση με λαθρεμπόριο ανθρώπων ή άλλα σχετικά. Εκεί υπάρχουν κάποιες τεχνικές πτυχές. Θα θυμίσω ότι μία βασική ιδέα πίσω από την πρότασή μας είναι και η προστασία των εξωτερικών συνόρων Σέγγεν. Δηλαδή, εάν μια χώρα μέλος που δρά μέσα στις επιχειρήσεις ε, Frontex έχει σχετικές ανησυχίες, δεν θα, είναι, δεν είναι δυνατόν οι υπόλοιποι να παραμείνουν με τα χέρια σταυρωμένα, εφόσον ανεπίτρεπτες είσοδοι μέσω του Frontex παρατηρούνται και βεβαίως και αυτό ισχύει και για τις αναθετήσεις είτε σε ε, εθνικά ύδατα είτε στα διεθνή ύδατα. Σε ό,τι αφορά τώρα την διαγραφή τμήματων για την αποβίβαση, ο κύριος Κοέλιο ανέπτυξε το θέμα. Δεν έχω πολλά να πω. Οι περισσότερε από τι διατάξει αυτέ περιλαμβάνονται στην ισχύουσα απόφαση του Συμβουλίου του 2010 και εφαρμόζονται στην πράξη. Το feedback που διαθέτουμε τώρα ομόφωνα από τι χώρε μέλη είναι ότι οι διατάξει αυτέ λειτουργούν καλά και δεν προκαλούν προβλήματα. Το ερώτημα άρα εδώ δεν είναι αν χρειάζονται ή όχι, αλλά αν ίσω πρέπει να ε, μπει σε περισσότερε λεπτομέρειε ω συνομοθέτη. Τελευταίο θέμα, τροπολογίε για ενδεχόμενε διμερεί συμφωνίε μεταξύ χωρών μελών και τρίτων χωρών. Ασφαλώς μπορούν να γίνουν αυτές οι διασταυρούμενε παραπομπές εφόσον το επιθυμείτε. Βασική αρχή ωστόσο είναι ότι οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού υπερισχύουν πάνω σε αυτές τις, ε, απέναντι σε αυτές τις διμερείς συμφωνίες. Ευχαριστώ που ήσασταν και σύντομος η κυρία Βέρση που είναι εκπρόσωπος της Λιθανικής Προεδρίας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε. Και εσείς κύριε Σιγητά και εσείς μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ανάλυση που κάνει η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου της πρότασης αυτής μετά από την απόφαση του δικαστηρίου. ότι οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις πρέπει να εγκριθούν μέσα σε μια εύλογη προθεσμία. Ε, η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου έχει εγκύψει τη μελέτη της πρότασης. Υπάρχει η ειδική ομάδα εργασίας του Συμβουλίου που είναι αρμοδία για την πρόταση. Έχουμε παραπέμψει το θέμα βέβαια και στην Επιτροπή Μετανάστευσης και Συνόρων που είναι υψηλού επίπεδου. Η ιδέα επιτροπή αυτή υψηλού επίπεδου έχει συζητήσει τα άρθρα 9 και 10. Αυτό δεν συνέβη στις 22 Δεκάτου. Νέα συμβαστική πρόταση έχει εκπονηθεί, η οποία θα συζητηθεί στις 22 Ενδεκάτου στην Ομάδα Εργασίας Συνόρων και εφόσον η έκβαση εκεί είναι θετική, θα διαβιβάσουμε την πρόταση σε άλλα όργανα του Συμβουλίου θα ήθελα επίσης με την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το επιτυχές έργο του στην Επιτροπή σας και βεβαίως είμαστε διατεθειμένες να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τον εισηγητή και να σας ενημερώνουμε για την πρόοδο της προτάσεως στο Συμβούλιο. Επίσης, επιθυμούμε να συνεργαστούμε με σας σε πνεύμα συνεργασία και σεβασμού. σεβασμού. Ευχαριστώ. Οι σκιώδει εισηγητέ τώρα. Εκτός από τους σκιώδει εισηγητέ, έχω δύο αιτήσει παρεμβάσεων. Ματιέ Κορατσαμπίλτ. Άλλος κανείς, εσείς ναι, σύμφωνοι. Α, και ο κύριος Ιακολίνο. Και ο κύριος Μπρον. Άρα μπορώ να κλείσω τον κατάλογο των αγορητών. Κύριε Βάιντεν Χόλτσερ. Ευχαριστώ να ξανασκεφτούμε κατά βάση το ότι εδώ δεν πάμε να ρυθμίσουμε την πρόσβαση στην Ευρώπη. Έχουμε μια κατάσταση στην Μεσόγειο που είναι κατάσταση έκτακτη. Με κανένα τρόπο βεβαίως δεν μπορεί να αποτελέσει την συνήθη πρόσβαση στην Ευρώπη. Αυτά που βλέπουμε εκεί είναι ε, καταστάσεις έκτακτες, τραγικές και η λύση του προβλήματος δεν μπορεί να περάσει μέσα από αυτήν την οδηγία. Πρόκειται για τελείως διαφορετικά πράγματα, τα οποία πρέπει να λυθούν στα πλαίσια της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Εκεί πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο βεβαίως. Εδώ το επιδιωκόμενο είναι να εφαρμοστεί η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον εισηγητή που έλαβε ξεκάθαρη θέση και δεν έχουμε και άλλη δυνατότητα παρά να προχωρήσουμε στη ρύθμιση αυτή. Υπάρχει βεβαίω αυτή η ευρωπαϊκή αρμοδιότητα και η ιδιαίτερα ευγνώμων που αυτή την γνώμη προβάλλει τόσο σαφώς ο ε, εισηγητής. Άλλωστε την συμμεριζόμαστε οι περισσότεροι εξημών. Για τη ρύθμιση των προβλημάτων αυτών στην Μεσόγειο έχουν να Δεν είναι δυνατόν αυτή η κοιτίδα του πολιτισμού να γίνει πια ο τάφος του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Είναι πράγματα απολύτως απαράδεκτα αυτά που συμβαίνουν εκεί. Πρέπει να κάνουμε κάθε τι το δυνατό για να αποτρέψουμε τέτοιες τραγωδίες. Με την έννοια αυτή θεωρώ ότι πρέπει να αποδώσουμε τα ίδια δικαιώματα στους ανθρώπους αυτούς που περνούν από τις θάλασσες όπως σε αυτούς που έρχονται μέσα από τα χερσαία σύνορα. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι διασώζονται από ναυάγια πρέπει να έχουν το δικαίωμα του διερμηνέα να ακουστούν και ούτω καθεξής. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει διακριτική μεταχείριση σε βάρος τους. Γι' αυτό υποστηρίζω όλες τις τροπολογίες που κινούνται στην κατεύθυνση αυτή. Και η απαγόρευση επανεισδοχής είναι εν προκειμένου σημαντική. Δεν μπορούν να είναι pushback, δεν μπορούμε δηλαδή να τους σπρώξουμε να πάνε πίσω διότι αυτό αντιβαίνει στην ε, υποχρέωση εξέτασης των ετοιμάτων του ατόμου. Αυτή είναι η γραμμή του συγητή και με βρίσκει σύμφωνο. Και είναι σημαντικό αυτό να εκφραστεί και μέσα από τις τροπολογίες. Να αποτραπούν αυτά τα pushback τα οποία είναι ε, απολύτως ε, ανάρμοστα με την ε, προσπάθεια προστασίας των δικαιωμάτων του ατόμου. Η κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή για τη λεπτομερή παρουσίαση. Θέλω να αναφερθώ σε τρία σημεία σχετικά με την έκθεση αυτή. Καταρχήν ε, το θέμα της έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε ότι αν δεν έχουμε πλήρες κανόνες δεν μπορεί να είναι και δεσμευτικοί κανόνες για την έρευνα και διάσωση. Επομένως, πιστεύω πως δεν πρέπει να δεχτούμε τις τροπολογίες του κ. Δίας Δεμέρα που βασικά θα σήμαιναν διαγραφή του άρθρου 9 για την έρευνα και διάσωση. Νομίζω ότι υποσκάπτει αυτό το στόχο μας να έχουμε δεσμευτικού κανόνες για το να σώσουμε τη ζωή στη θάλασσα. Επίσης πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να διατηρήσουμε στους ορισμούς ε, το τι σημαίνει να βρίσκεται κάποιος σε αυτή τη δύσκολη θέση. Δηλαδή ποιος πρέπει να διασώζεται Έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που πεθαίνουν στη Μεσογείο. Θέλω να αναφέρω το τι έγινε το 2011 με 72 ανθρώπους που ζητούσαν να διασωθούν ε, και έστειλαν σήμα κινδύνου, αλλά είπαν ε, τα κράτη, οι αρχές του κράτους μέλους ότι δεν κατάλαβαν ότι πρόκειται για επίγον κλείσει επίγουσα κλίση κινδύνου και έσωσαν μόνο 9 ανθρώπου τελικά. Έτσι λοιπόν, εγώ νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει να έχουμε μια κατάσταση κινδύνου. Έτσι λοιπόν, εγώ θα σας παροτρύνω να μην δεχτείτε καμία διαγραφή αυτών των ορισμών. σε σχέση με το κίνδυνο και ε, το συναγερμό. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό αν θέλουμε να έχουμε πρόοδο στο θέμα της διάσωσης της ζωής στη θάλασσα. Επίσης, δεν νομίζω ότι πρέπει να πέσουμε στην παγίδα που έχουν στήσει τα κράτη-μέλη της Νότιας Ευρώπης, γιατί μετά την ε, Λαπεντούζα και ο κύριος Σαλφάνο είπε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη και θέλουμε μεγαλύτερη βοήθεια από την Ευρώπη, αλλά τελικά όταν ε, έχουμε κοινέ επιχειρήσεις από τη Frontex και έχουμε κανόνες, τότε η Ιταλία και άλλα κράτη-μέλη δεν συμφωνούν. Και τώρα σε ό,τι αφορά το pushback, την απόφυση ε, να θυμόμαστε την απόφαση του δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να ενημερώνουν οι διασωθέντες για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για να μην αποβιβάζονται σε τρίτες χώρες. Θα πρέπει να έχουν πρόσβαση και σε προσφυγή επίσης ε, αποτελεσματική προσφυγή. Επίσης, ε, ε, και οι συνοριοφύλακες θα πρέπει ε, πάντοτε να εξετάζουν τις προσωπικές καταστάσεις, τις προσωπικές συνθήκες στις οποίες βρίσκεται ο μετανάστης και να επιτελούν τα καθήκοντά τους. Αυτά τα είπε το δικαστήριο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η απόφαση αυτή πρέπει να εφαρμοστεί και επομένω η πρόταση τη Κομισιόν δεν σέβεται την απόφαση. Δεν αρκεί να ενημερώνονται οι άνθρωποι ότι θα αποβαστούν σε ένα συγκεκριμένο μέρο, αλλά πρέπει να ενημερώνονται τι μπορούν να κάνουν κατά αυτού και να τους δίνονται οι δυνατότητες να αποφεύγεται αυτή η αποβίβαση. Και εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι δυνατό αυτό επί του σκάφους, γιατί δεν μπορείς να έχεις μια σειρά νομικών και διερμηνέων επί του σκάφους. Εγώ νομίζω ότι αυτά τα pushbacks, αυτές οι αποθήσεις ε, μπορούν ε, να αποφευχθούν και ε, κανένας κανόνας δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην ανοιχτή θάλασσα. Θα πρέπει να αποβιβάζονται οι άνθρωποι αυτοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου θα έχουν μία δίκαιη διαδικασία και μία δίκαιη δίκη. Όμως φαίνεται ότι υπάρχουν εδώ κάποιοι που πιστεύουν ότι μπορεί να γίνεται αυτό στην ανοιχτή θάλασσα αλλά εγώ νομίζω ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο και τέλος, συγγνώμη που θα πρέπει να ευθυγραμμίσουμε την νομοθεσία μας με το πρωτόκολλο κατά της ελευθερμπορίας μεταναστών, γιατί και εδώ ε, μιλάμε για πρέπει να συλλαμβάνουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι δουλέμποροι και όχι να συλλαμβάνουμε ανθρώπους που είναι μετανάστες. Μάλιστα, συγγνώμη που σας διακόπτω μερικές φορές, λέει Πρόεδρος, αλλά νομίζω ότι για να είναι ε, η συζήτηση εδώ ζωντανή ε, και για να σεβόμαστε και τους άλλους συναδέλφους πρέπει να περιοριζόμαστε στα τρία λεπτά. Κυρία Έρνστ. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω πως η πρόταση του κύριου Κόελιο έχει πραγματικά μία μεγάλη δυνατότητα, δίνει μια μεγάλη ευκαιρία για να επέλθει τάξη και βελτίωση για τους ε, μετανάστες. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή που έχουμε εδώ και ξέρω πως δεν μπορούμε να λύσουμε το μεταναστευτικό πρόβλημα. Είναι σαφές αυτό, ε, όπως είπε και η προηγούμενη μιλήτρα και οι προηγούμενοι συνομιλητές μου έτσι κι αλλιώς. Ε, το θέμα όμως ε, είναι το πώς αντιμετωπίζουμε την μετανάστευση και πιστεύω πως πραγματικά έχει ο συνάδελφος καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να έχει ένα ισορροπημένο κείμενο. Εγώ στηρίζω την πρόταση αυτή. Πιστεύω πως δεν μπορεί με κανένα τρόπο να είναι αποδεκτή αυτή η διαδικασία έτσι όπως γίνεται τώρα. Ε, χρήζουν διεθνούς προστασίες αυτοί οι μετανάστες και ε, δεν πρέπει να τιμωρούνται. Πρέπει να γνωρίζουμε την ε, νομική βάση επίσης σε ορισμένα κράτη-μέλη για τους ε, μετανάστες αυτούς και υπάρχει διαφοροποίηση για παράδειγμα μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων και αυτό αυτή τη στιγμή ε, πρέπει να το εξετάσουμε και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να, θέτεται, να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή των ανθρώπων αυτών. Χρειαζόμαστε μια δυνατότητα ύπαρξης νομικών μέσων, ε, τα οποία να είναι στη διάθεση των μεταναστών. Είναι πραγματικά, και το ξαναλέω αυτό, μία ευκαιρία και απευθύνομαι και στο Συμβούλιο και θα ήθελα να σας πω ότι πραγματικά αυτό που μας λέτε δεν είναι τοποθέτηση. Δεν, δεν σημαίνει τίποτα το ότι έχετε δημιουργήσει μία ομάδα εργασίας. Στηρίζω πολύ τον κύριο Κοέλιο, ιδιαίτερα στο σημείο όπου αναφέρεται για ε, το ποιο έχει την αρμοδιότητα να συζητήσει αυτό το πράγμα. Και σας παρακαλώ, ναι, αυτή είναι η δουλειά μας. Η δουλειά μας και ω και συζητητέ και είμαι σε πλήρη τιμότητα να συνεργαστώ απόλυτα μαζί σας. Αλλά πραγματικά θεωρώ πολύ προβληματική τη στάση αυτών των έξι κρατών μελών και σκεφτείτε ότι του χρόνου έχουμε ευρωεκλογέ και πραγματικά ε, αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση βλάπτουν τη, τη φήμη μας, την καλή μας εφήμη. Γι' αυτό σας παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι ευρωβουλευτές, ε, πρέπει να πάρετε τα πράγματα στα σοβαρά. Υπάρχει ανάγκη, εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές και δεν έχει καμία σημασία αν κάποιος είναι μετανάστης ή όχι, είναι άνθρωπος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, τώρα θα δώσω το λόγο και στα άλλα μέλη που ζήτησαν το λόγο. Έχω τέσσερις ομιλητές στον κατάλογο. Σας ζητώ να κρατήσετε το όριο των τριών λεπτών. Η κυρία Ματιέ, η κυρία Κοράτσα Μπίλτ, ο κύριος Ιακολίνο και ο κύριος Μπρόντς. Κυρία Ματιέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το εξαιρετικό του έργο και τους κοιόδες εισηγητές που ενέσκυψαν εις βάθος το ζήτημα. Τώρα, ο αριθμός των τροπολογιών που εξετάζουμε σήμερα μας δείχνουν ότι πρέπει να κάνουμε πολλά ακόμα για να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση του Κοινοβουλίου για το κείμενο αυτό. Και θα ήθελα να επιμείνω στο σημείο αυτό. Κανείς ε, εδώ δεν είναι κατά της διάσωσης στη θάλασσα. Και φυσικά όλοι συμφωνούν για να πούν αν ένας άνθρωπος είναι σε κίνδυνο, αν ε, όταν περνά από μια τρίτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κινδυνεύει από πνιγμό, Φυσικά πρέπει να σώσουμε το άτομο αυτό αν κινδυνεύει η ζωή του και φυσικά και όλες οι διεθνείς συμφωνίες προβλέπουν τη διάσωση αυτού του αντόμου. Και φυσικά όλοι συμφωνούν σε κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι κάποιος στο Κοινοβούλιο αμφισβητεί αυτό το θέμα. Όμως το θέμα δεν είναι εδώ σήμερα. Το ερώτημά μου αφορά περισσότερο την πρακτική και την νομική σκοπιά. Είμαστε αρμόδιοι για ε, να νομοθετήσουμε δεσμευτικά για το θέμα της διάσωσης στη θάλασσα. Ήδη έχουμε διεθνές δίκαιο για το θέμα αυτό. Έχουμε τη Διεθνή Σύμβαση για την έρευνα και τη διάσωση στη θάλασσα προβλέπεται ήδη υποχρέωση να προσφέρεται βοήθεια στα άτομα σε κίνδυνο, όποια και είναι η εθνικότητά του ή το καθεστώ του. Προβλέπεται να ιδρυθούν κέντρα συντονισμού, να υπάρχει επιμερισμό των ζωνών μεταξύ τη αστυνομία, ανταλλαγή πληροφοριών ε, και να υπάρχουν και λεπτομερή σχέδια και τα έξι κράτη-μέλη έχουν κυρώσει αυτές τις διεθνείς συμφωνίες. Ε, Επομένως, σήμερα χρειαζόμαστε ένα νέο μέσο που προτείνεται από την Κομισιόν και θα δημιουργηθεί σύγχυση. Με αυτό, αν έχουμε ευρωπαϊκούς κανόνες ε, για το θέμα αυτό, με ένα νέο νομικό καθεστώς που θα εφαρμόζεται παράλληλα με τη διεθνή νομοθεσία, αυτό αναρωτιέμαι σήμερα. Δηλαδή πώς θα ξεχωρίσουν όσοι δραστηριοποιούνται επί τόπου την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία από την Εθνική Νομοθεσία γιατί όταν κάποιος πρέπει να διασώσει μία ζωή είναι ε, επίγον το ζήτημα. Θα μπορεί τότε να κάτσει να ξεχωρίσει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία από την Εθνική Νομοθεσία. Αυτό ανερωτιέμαι και επίση. Ε, θα ήθελα να σα πω ότι αυτό θα εφαρμοζόταν μόνο στι επιχειρήσει Frontex. Ε, δηλαδή, όταν κάποιο στα πλαίσια μια επιχείρησης Frontex θα εφαρμόσει κάποιους κανόνες, ενώ όταν έχουμε μια εθνική επιχείρηση θα πρέπει ο αρμόδιος να θυμάται και να εφαρμόζει άλλους ε, κανόνες. Ε, και μπορώ να σα πω ότι ε, μπορεί και κάποιοι να συμμετέχουν στην ίδια επιχείρηση και να πρέπει να εφαρμόσουν διαφορετικούς κανόνες. Θα υπάρχει σύγχυση λοιπόν μεταξύ της διεθνούς νομοθεσίας των ευρωπαϊκών κανόνων ε, για τα σκάφη που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις Frontex και για τα σκάφη που δεν συμμετέχουν. Και όλα αυτά θα γίνονται ενώ θα είναι κατεπίγουσα η ανάγκη γιατί θα μιλάμε ότι ε, το κλίμα θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο και θα βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν ε, εγώ νομίζω ότι αμφισβητού, πρέπει να αμφισβητήσουμε κάπω αυτή τη νέα πρόταση, γιατί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα φυστάμενα μέσα. Κυρία Κορατσαμπίλη, νομίζω ότι χρειαζόμαστε νέου κανόνε, όχι κοινού κανόνε για την ασφάλεια δικαίου. Αυτοί οι κοινοί κανόνε θα βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν καλύτερα την ε, υφιστάμενη διεθνή και ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν βλέπω να υπάρχει αντίφαση εδώ. Αντίθετα, μαζί με τη Eurosur και του κοινού κανόνες, από το 2010 Υπάρχει σχετική έκκληση. Εγώ πραγματικά υποστηρίζω τον κύριο Κοέλιο και την πρόταση της Κομισιόν να υιοθετηθούν αυτοί οι κανόνες εντός αυτής της θητείας. Ελπίζω να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το διέξοδο. Χρειαζόμαστε κοινού κανόνες για την έρευνα, τη διάσωση και τη σύλληψη, γιατί πρέπει να σώσουμε ζωές. Και βλέπουμε ότι το πρόβλημα είναι η ερμηνεία των κανόνων στην πραγματικότητα. Υπάρχει αβεβαιότητα στα κράτη-μέλη για το ποιο είναι υπεύθυνο να αναλάβει δράση. Και γι' αυτό αυτοί οι κοινοί κανόνε θα έπρεπε να ξεκαθαρίσουν ποιο είναι υπεύθυνο να αναλάβει δράση και πού. Πιστεύω ότι καταρχήν πρέπει να σώσουμε ζωές που πιστευω οτι καταρχην πρεπει να σωσουμε ζωε που ειναι το πιο σημαντικό, αλλά επίση πρέπει να βοηθήσουμε και τα κράτη-μέλη στα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, που νιώθουν αυτή την τεράστια πίεση. Επίσης νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο να καταπολεμηθεί το διασυνορικό έγκλημα και η εμπορία ανθρώπων. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε σοβαροί σε σχέση με το να αποτρέπουμε τραγωδίες όπως τις Λαμπεντούζα θα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα και να θετήσουμε αυτά τα μέτρα. Εγώ έχω καταθέσει κάποιες τροπολογίες για τα παιδιά, ελπίζω να με υποστηρίξετε γιατί φυσικά τα παιδιά και οι ασυνόδευτοι ανήλυτοι είναι οι πλέον ευάλωτοι από όσου φτάνουν στα θαλάσσια σύνορά και χρειάζονται βοήθεια συχνά και όταν είναι στη θάλασσα. Και έχω καταθέσει και μια τροπολογία σχετικά να το προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε αν υπάρχουν επί των σκαφών αυτών άνθρωποι που έχουν ιδιαίτερε ιατρικέ ανάγκε για να αξιολογήσουμε αν χρειάζεται ιατρική επέμβαση επιτόπου. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιακολίνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή όλες τις συνεισφορές των συναδέλφων για ένα ζήτημα ιδιαίτερα επίκαιρο και πολύ συγκεκριμένο. Αλλά είναι και ιδιαίτερα πολύπλοκο και ευχαριστώ τον εισηγητή, τον κύριο Κοέλιο που παρουσίασε αυτή την ε, ιδιαίτερα λεπτομερή έκθεση. Τώρα, θα ήθελα να κάνω κάποια συγκεκριμένα σχόλια και εγώ έχω καταθέσει μια σειρά τροπολογίων και πρέπει να πω δίνει μεγάλη έμφαση στο υπάρχει ειδική κατανομή των ζωνών της Frontex στη Μεσόγειο. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την επιχειρησιακή ικανότητα της Frontex και να εγγυηθούμε αυτή την έκτακτη συνεργασία σε μέσα και σε πόρους που είναι απαραίτητα για να αντιμετωπιστεί μια συνεχής κατάσταση κατεπίγουσα. Αναφερθήκατε κάποιοι συνάδελφοι και στη Λεμπεντούσα έχουν περάσει 40 μέρες ε, στις 3 Οκτωβρίου ε, χώρα. Η κυρία Μάστρομ και ο κύριο Μπαρόσο πήγαν στη Λεμπεντούσα και ανακοίνωσαν συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Εν τω μεταξύ ξεκίνησε η Ιταλία την επιχείρηση Mare Nostrum αλλά το μόνο κράτος που έδωσε μέσα είναι η Σλοβενία. Το λέω αυτό γιατί, όχι γιατί προέρχομαι από τη Σικελία και από την Ιταλία ε, κατ' επέκταση, αλλά και για άλλο λόγο, γιατί, κυρία Ματιέ, πρέπει να δούμε τι συμβαίνει συγκεκριμένα, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Σας δούμε τώρα τι συγκεκριμένες δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Κάρλος με τον μπλοκ των έξι χωρών, με τον μπλοκάρισμα των έξι χωρών. Ε, των ε, ερευνών και της διάσωσης. Εγώ νομίζω ότι αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά να τα δούμε και στα πλαίσια των συμφωνιών που θα υπογράψουμε με τις τρίτες χώρες. Ε, και επίσης κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι ο συντονισμός μεταξύ του Διεθνούς Κέντρου και των Εθνικών Κέντρων για να έχουμε αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Ας επανέλθουμε τώρα στο πιο επίμαχο θέμα. Εμείς θα πρέπει να έχουμε μια κοινή προσέγγιση σε ό,τι φορά τη μεταναστευτική πολιτική, το δικαίωμα του ασύλου, μια προσέγγιση που θα βασίζεται στην ευθύνη και στην αλληλεγγύη των κρατών μελών. Αλλά επί του συγκεκριμένου, αν πρέπει να διαφοροποιήσουμε τις επιχειρήσεις που γενικά διέπονται από το διεθνές δίκαιο, από τις επιχειρήσεις ε, που βρίσκονται υπό την αιγίδα της Frontex, θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε αντικειμενικές δυσκολίες και φυσικά πρέπει να βρούμε ένα σημείο ισορροπίας, αλλά είναι αλήθεια ότι και οι επιχειρήσεις της Frontex αποτελούν ε, ουσιαστικά ένα πολύ μικρό αριθμό επιχειρήσεων σε σχέση με τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν μένα τα κράτη, με η Ελλάδα, η Μάλτα, η Κύπρος, η Ιταλία, μόνες τους πρέπει να στηρίξουν αυτές τις ε, επιχειρήσεις. Έτσι λοιπόν ε, μπορεί λοιπόν, να υπερισχύει η λογική του να έχουμε μία προσέγγιση προς το διεθνές δίκαιο και εγώ εμπιστεύομαι τους συναδέλφους για να βρούμε ένα σημείο ισορροπίας και να ξεπεράσουμε αυτή την μειοψηφία ανάσχεσης. Γιατί θα πρέπει να προβούμε σε έρευνα και διάσωση στη θάλασσα, στα εγχωρίδια του κάθε κράτους μέλους. Μάλιστα, ευχαριστώ κύριος Μπρόνς. <clears throat> Ευχαριστώ. Ο κανονισμός τροποποιεί τις ρυθμίσεις για την διάσωση από μη δεσμευτικέ και τις κάνει δεσμευτικέ. Είναι προφανές ότι άνθρωποι που βρίσκονται σε κίνδυνο πρέπει να διασώζονται. Δεν το αμφισβητεί κανεί αυτό. Οι χώρε μέλη, μάλιστα, δεν χρειάζεται να του το πει κανεί αυτό, ή τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να χρειάζεται να του το πει κανεί αυτό. Ωστόσο, το πεδίο εφαρμογή διευρύνεται ώστε να περιλάβει και κανόνες για την αποβίβαση, δηλαδή που θα πρέπει να αποβιβαστούν τα πρόσωπα αυτά. Αυτό όμως είναι θέμα αρμοδιότητας των χωρών μελών υπό την επιφύλαξη των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η αιτιολογική έκθεση λέει ότι η ανάγκη προστασίας των συνόρων δεν πρέπει να αποβεί σε βάρος των ανθρώπινων δικαιωμάτων των μεταναστών. Όμως η αρχή της μη επανεισδοχής και οι αποφάσεις του δικαστηρίου, μήπως αυτές είναι καταστροφικές για την ε, δυνατότητα προστασίας των εξωτερικών συνόρων. Διότι αυτά σημαίνουν ότι οι ενδεχόμενοι αυτοί μεταναστές αρκεί να αποδείξουν ότι προέρχονται από επικίνδυνες χώρες είτε με χαρτιά είτε χωρίς για να τους δοθεί άσυλο. Η λειτουργία του, της αρχής ε, της μη επαναπροώθησης η αρχή αυτή είναι άμεσα υπεύθυνη για τις τραγικές τραγωδίες μάλλον που διευθυνθήκαν στη Μεσόγειο. Ευχαριστώ. Εδώ ολοκληρώνω τη συζήτηση και έτσι οδηγούμεθα και πάλι στον ε, εισηγητή. Κύριε εισηγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια που είπαν οι συνάδελφοι για την έκθεσή μου και στη κοινή προσπάθεια να βρεθούν λύσεις. Ευχαριστώ επίσης την Προεδρία του Συμβουλίου για τα καλά λόγια που είπε και για τις προσπάθειες που αναλαμβάνει και την πίεση που ασκεί στις χώρες μέλη ε, που διστάζουν για να λάβει την εντολή για τις διαπραγματεύσεις όσο δε τον συντομότερο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πρόταση συμβιβασμού δεν προβλέπει την διαγραφή των άρθρων 9 και 10 και κατά τη γνώμη μου αυτό ήδη είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Για να είμαι σαφής, παρακαλώ, για δύο λεπτά, Πρόεδρε. Γιατί τονίζω την ανάγκη να υιοθετηθούν τα 9 και 10. Γιατί δεν κατανοώ τις χώρες εκείνες οι οποίες επιθυμούν να διαγράψουν τα άρθρα αυτά. Διότι στην απόφαση του Συμβουλίου που ελήφθη με ομοφωνία τα άρθρα αυτά περιλαμβάνονταν είναι αλήθεια βέβαια ότι δεν ήταν δεσμευτικά, όμως υπήρχαν μέσα στην απόφαση. Κανείς στο Συμβούλιο, όταν ενέκριναν την απόφαση ομόφωνα, δεν είπε ότι δεν είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Συμφώνησαν. Τώρα η Κομισιόν μας προτείνει δεσμευτική απόφαση και κατά τη γνώμη μας και γνώμη μου θα πρέπει να υποστηρίξουμε την πρωτοβουλία της Κομισιόν Ίσως τώρα κάποιο θεωρεί ότι δεν είναι στην αρμοδιότητά μας. Το πολιτικό ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Μετά τα, όσα, μετά τα όσα συνέβησαν στην Μεσόγειο, όλοι στο Συμβούλιο, όλοι οι πρωθυπουργοί, όλοι οι αρχηγοί κρατών, είπαν να το σταματήσουμε. Αυτές, να σταματήσουμε τις τραγωδίες αυτές και γνωρίζω ότι πολλές αποφάσεις θα χρειαστεί να ληφθούν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Όμως, το πρώτο νομοθέτημα που έχουμε είναι αυτό. Τι πάμε να κάνουμε λοιπόν στο πρώτο αυτό νομοθέτημα. Θα παραστήσουμε ότι δίθεν η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει τίποτε και ότι μόνο οι χώρες μέλη οφείλουν να λάβουν τις αποφάσεις. Όχι. Όχι, δεν είναι προφανής η απάντηση αυτή. Όταν όλοι ζητούν περισσότερη Ευρώπη, θα πρέπει να δοθεί μια ευρωπαϊκή απάντηση. Και παρά το γεγονός ότι έχω κατανόηση για πολλές από τις τροπολογίες συναδέλφων μου, που θέλουν να πάνε ακόμα μακρύτερα, οφείλω τόσο να τους πω με την ίδια σαφήνεια ότι δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στις χώρες μέλη πράγματα τα οποία είναι καθαρά εθνικής αρμοδιότητας. Θα πρέπει λοιπόν να κρατήσουμε μια θέση ισορροπίας που κατά τη γνώμη μου έγκυται στο εξής. Ό,τι είναι ευρωπαϊκή επιχειρησιακή δράση Frontex θα πρέπει να υπάγεται σε ευρωπαϊκούς κανόνες. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε περαιτέρω, να ανοίξουμε συζήτηση δηλαδή με το Συμβούλιο γιατί ξεπερνούμε τις αρμοδιότητές μας και αναγκάζουμε τις χώρες μέλη να εκχωρήσουν κυριαρχία. Με τις συμβαστικές τροπολογίες που θα προτείνω θα εμείνω σε αυτή την ιδέα. Θα χρειαστεί να έχουμε δηλαδή περισσότερη Ευρώπη σεβόμενοι ταυτόχρονα τη νομική μας βάση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση αυτή. Θα διακόψουμε για λίγα λεπτά, διότι η ψηφοφορία προβλέπεται για τις 12 και 20 και ίσως ε, έλθουν και άλλα μέλη της Επιτροπής ε, στην ακριβή ώρα που προβλέπεται.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 Okay, please take your seats. going to... Αγαπητοί συνάδελφοι, να περάσουμε στην μόνη ψηφοφορία που έχουμε σήμερα το πρωί για την οδηγία για τους εποχικούς εργαζομένους. Ο κύριος Κλοντ Μωράς είναι εισηγητής. Όπως ε, παρουσιάστηκε από τον εισηγητή στην περασμένη συνεδρίαση, είχαμε βίτευξη συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση και η Επιτροπή Απασχόλησης ψήφισε σήμερα το πρωί επί το αποτελέσματο των διαπραγματεύσεων σε ό,τι αφορά τα τμήματα για τα οποία έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα και μου είπαν ότι υποστήριξαν τη συμφωνία. Ο εισηγητής προτείνει να ψηφίσουμε το συμβιβαστικό κείμενο σε μπλοκ. Είστε όλοι έτοιμοι λοιπόν για την ψηφοφορία. Πολύ ωραία. Θα έχουμε λοιπόν μία και μόνη ψηφοφορία επί του συμβιβαστικού κειμένου, έτσι όπως προτείνεται από τον εισηγητή. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Σαφής πλειοψηφία. Και περνάμε μέσω στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική. Άρχεται η ψηφοφορία. δεν έχετε κάρτα, θα μετρήσουμε την ψήφο σας. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Εκτός από το Γιάνν, πέρας. Μάλιστα, μια πολύ καλή πλειοψηφία μαζί με το Γιάνν, 33 ψήφοι υπέρ. Συγχαρητηρία στον εισηγητή. Και ερχόμαστε στο τέλος της σημερινής μας συνεδρίασης. Να υπενθυμίσω σας παρακαλώ, ένα λεπτό. Το απόγευμα θα συνεδριάσουμε στην αίθουσα 2Q2. Σας ευχαριστώ και θα τα πούμε το απόγευμα.